Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ιδάλω δεν θα προλάβουμε στο ωράριο που προβλέπετε. Στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται το σημείο 15. Στα πλαίσια της έκθεσης Μερκαστέλο για το πρόγραμμα προς τους πλέον μενεκτούντες. Έχουμε οργανώσει δημόσια ακρόαση με αρκετούς ε, παρεμβαίνοντες, πέντε. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερως που βρίσκονται μαζί μας και νομίζω είναι σημαντικό να ακούσουμε για τις δικές σας μαρτυρίες και τεχνικές γνώσεις. Δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι για να παρουσιάσετε τι δικέ σα ε, παρατηρήσει. Έχετε περίπου 5 λεπτά στη διάθεσή σα. Πριν όμως σα δώσω το λόγο, να δώσω το λόγο στην κυρία Έμπλερ Κοστέλο για να τοποθετηθεί αρχικά και να σας καλέσει να αποκριθείτε ουσιαστικά σε αυτά τα οποία έχει ανάγκη να γνωρίζει και η Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο, κυρία Συγκήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες καθώς και όσους βρίσκονται σε αυτήν την ε, ακρόαση. Το πρόγραμμα FEED, το επιστημιστική βοήθεια, βοήθεια μάλλον ευρωπαϊκή βοήθεια για τους πλέον μενεκτώντες, είναι ένα ε, σημαντικό θέμα που απασχολεί την Επιτροπή μα. 116 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγονται την κατηγορία των πλέον μεονεκτούντων, μεταξύ των οποίων και άστεγοι. Εδώ υπάρχει πρόταση για ένα νέο ταμείο. Το Ταμείο για την και Βοήθεια, το Ταμείο Φίντο, όπω έχει ονομαστεί, και η προτινόμενη πρικοδότηση ήταν αρχικά 2,5 δις αλλά τώρα έχει κατέβει στα 2,1 δις ευρώ. Ο στόχος αυτής της ακρόασης είναι να συναντήσουμε εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όπως είπε και ο Πρόεδρός μας, να ακούσουμε τις δικές τους απόψεις για την πρόταση εδώ για την πρόταση του Ταμείου ΦΙΔ. Αυτή είναι η δική μας προσπάθεια. Ξέρω ότι είναι πολλέ οι με κυβερνητικέ οργανώσει που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, γι' αυτό έχουμε και τόσε παρεμβάσει σήμερα εδώ. Λυπούμε που δεν μπορούσαν βέβαια να παρέμβουν κι άλλοι, όσοι ήθελαν να συνεισφέρουν στη σημερινή ακρόαση. όμω ο κατάλογο των παρεμβαινόντων όπω τον βλέπουμε νομίζω ότι κατοπτρίζει και τι προτεραιότητε μα, αυτέ που απεικονίζονται στην πρόταση FID, που ασχολούνται με την στέγαση, τη σύντηση, ε, την βοήθεια για τα παιδιά επίσης που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία των πλέον μειονεκτούντων. Είναι μεγάλη χαρά μας λοιπόν να μπορούμε να συναντήσουμε σήμερα τους ε, συμμετέχοντες και να συζητήσουμε μαζί τους. Από τους οργανισμούς που παρίστανται θέλουμε να δούμε κατά πόσον στην σημερινή τους ε, δουλειά και στην σημερινή γνώση του προγράμματος όπως την έχουν αποκομίσει κατά πόσον έχουν εντοπίσει σημεία, προτάσεις, συστάσεις για βελτιώσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα θέλαμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τους ε, παρεμβαίνοντες που ήρθαν σήμερα εδώ. Και βεβαίως ευχαριστούμε και όσους υπο... τους υπόλοιπους που ενδιαφέρθηκαν για το θέμα αυτό, παρόλο που μπορεί να μην μπόρεσαν να παρέμβουν ή να παραστούν. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τη συνεισφορά των ε, ομιλητών. Πρόεδρος, ευχαριστώ να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Μπέρτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης των Ρεστών Ντικέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα πρώτα, θα σας πω για δύο, αυτό το πρόγραμμα της βοήθειας, τι μας επιτρέψουμε να κάνουμε θα πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί προσπαθείτε πριν αποφασίσετε να καταλάβετε, να ακούσετε αυτούς που δουλεύουν ε, επί τόπου. Τους μάχημους. Πάρα πολύ ενθαρρυντικά είναι όλα αυτά. Είχαμε και την επίσκεψη Μπαρόσο στην Επιστήμη Τράπεζα, κ. Αντόρ. Τους ε, υποδέχτηκα ε, τον Νοέμβριο. Κυρία Κοστέλο, κυρία Μπερές, για να δούμε τις δραστηριότητες μας. Για να δουν τι κάνουμε. Οπότε έχουμε ξεκινήσει από το 1987 αυτό το πρόγραμμα και είμαι θελοντής από το 1986 και από, ήξερα την κατάσταση πριν και μετά το πρόγραμμα. Γίνεται μεγάλη διαφορά γιατί έχουμε κάποιες σταθερές εισφορές, έχουμε πολλά είδη πρώτης ανάγκες που δίνονται, οπότε και γι' αυτό ο φορέας μας μπορεί τώρα να κάνει μια ισόρροπη τακτή ε, δράση, να τη συνεχίσει, να καταπολεμήσουμε την έλλειψη των τροφίμων, ε, την κοινωνική ένταξη και να βοηθήσουμε να μην ε, διασπαθίζονται τα τρόφιμα. Και μαζεύαμε αυτό το οποίο οι άλλοι δεν ήθελαν. Ο καθένας έδινε όσο ήθελε Όποιο ερχόταν εδώ πέρα και οπότε για αυτό το λόγο προσπαθούσαμε να συνεργαστούμε με τους ε, θελοντές οι οποίοι είναι σημαντικό τμήμα ε, μαζεύουν χρήματα, τρόφιμα και οπότε από τότε που αυτό το πρόγραμμα υπάρχει άλλαξε πως καλύτερη κατάσταση ο φορέας του οποίου προεδρεύω έχουμε 15 εκατομμύρια ε, και 86, ε, εκατομμύρια κόσμο τρέφουμε και προσπαθούμε έτσι να βοηθήσουμε και για τη δουλειά, βοηθούμε για στέγαση, έχουμε μικροπιστώσεις ε, πολιτιστικά, βοηθάμε για το σχολείο, κατά του αναφαβητισμού για δεκάδες χιλιάδες πρόσωπα και αποδίδω σύστημα διότι έχουμε, έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι πολλές φορές έρχονται τη μία χρονιά, δεν έρχονται την επόμενη γιατί η κατάσταση τους έχει, έχει βελτιωθεί. Το 45% αυτόν βοηθάμε. Έχουμε 18 εκατομμύρια Ευρωπαίων οι οποίοι βοηθούνται από το πρόγραμμα και αυτό είναι ένα από τους βασικούς στόχους είναι βασικός στόχος ένταξης και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτούς που είναι οι, πιο μειονεκτούντες, οι πιο φτωχοί, που δεν τους καλύπτει κανένα πρόβλημα, πρόγραμμα. Και αυτό γίνεται με τρόπο τακτό για όλες αυτές τις φάσεις και ε, προσπαθεί ε, για το, το, το κράτος να βοηθήσει Έχουμε το ελεγκτικό συνέδριο της Γαλλίας που έκανε μια έρευνα και είπε ότι ε, δίνουμε 5% ε, περισσότερα από όσο δίναμε πριν και έχουμε και κάποιες επιδοτήσεις. Εάν το πρόγραμμα αυτό δεν περάσει, εάν αυτό το ποσό συρρυκνωθεί, τότε δεν θα έχουμε αρκετά χρήματα σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Αυτό είναι βέβαιο και στην Ευρώπη η, κοινωνική συνοχή συνέχεια επιδεινώνεται. Θα υπάρχουν πάρα πολύ βασικές συνέπειες για την διατροφή, για την κοινωνία, ε, καταστάσεις ακραίες φτώχειας και θα υπάρχουν και οικολογικές συνέπειες όσον αφορά την διασπάθηση των τροφίμων, πρόβλημα με την ασφάλεια, με τη σταθερότητα σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιοχές, γιατί ότι όταν, όταν δεν υπάρχει ανθρωπινός, η ανθρωπιά τότε έχουμε άλλους ε, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ε, αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε, σε μειονεκτούσα θέση. Άρα αυτό θα μαυρώσει την εικόνα της Ευρώπης, την ε, αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία της Ευρώπης. Αυτό για το οποίο πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση το, τον Νόμπελ. Κρίση οικονομική, παροξισμός και Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το κοινωνικό ταμείο. Αλλιώ είναι η κατάσταση παράλογη. Τα, αυτά τα εστιατόρια της καρδιάς τα ξεκίνησε ο Κολλού και είχε ασχοληθεί και ο ίδιος ο ζακτελόρο πρόεδρος και είπαμε, αντί να γίνεται αποθήκευση των παραπάνω τροφίμων να μοιράζονται. Είδατε πόσο ε, συναισθηματικό, πόσο φορτισμένος είμαι για αυτό το πρόγραμμα και επομένως θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει το Συμβούλιο. Αν δεν ψηφιστεί το πρόγραμμα, δεν θα έχουμε ενέργεια, δεν θα έχουμε τους πόρους, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε αυτή την κρίση που έχει πλήξει όλα τα κράτη. Τους μετανάστες, τους ξένους και τους ντόπιου σε κάθε κράτος. Και πριν και μετά. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι το Κοινοβούλιο να βοηθήσει να έχουμε τα μέσα για να κατολίσουμε τη φτώχεια, την κοινωνική ένταξη κατά του κοινωνικού αποκλεισμού όλων. Πρόεδρο, και τώρα παρακαλώ οι άλλοι ομιλητές να σεβαστούν το χρονικό όριο, να μιλάνε πιο αργά και... Και μην ξεχνάτε ότι ο σκοπός είναι να μας βοηθήσετε στο έργο μα ω νομοθέτε. και να δούμε τι θα γίνει με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί επί τη βάση αυτού του, ταμείου αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε. Έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής. Και έχουμε βέβαια αυτή την παρεμποδισμία ψηφία στο Συμβούλιο για αυτό το πρόγραμμα. Εδώ δεν έχουμε πάντω κάποιου που θέλουν να πανεμπούν στο και αν που είχαμε είναι καλά ε, κρυμμένοι. Οπότε έτσι να δουλέψουμε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι θα αποδώσει αυτή η ακρόαση. Έτσι θα μας βοηθήσετε. Είτε σας αρέσει είτε όχι το κείμενο. Μας δεν το πράγμα είναι σημαντικό, το ξέρουμε. Όχι, όχι, δεν το λέω κατά του Ολιβιέ Μπερτά. Το λέω για να έχει αποτελεσματικότητα η, η ακρόασή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Λέω κύριος Φάρελ. Αυτό το πρόγραμμα να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Μια έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια στα πλαίσια Τη πρόταση που τώρα συζητείτε, Τη πρόταση τη Κομισιόν. Δουλεύουμε με την Φιάνσα, τον Ερυθρό Σταυρό, τον, την Κάριτας και άλλε οργανώσεις στην Ευρώπη και έχουμε πάρα πολύ σημαντικέ ε, εμπειρίε. Όλα αυτά τα οποία εδώ θα ακούσουμε στην εκρόαση. Και πρώτα πρώτα πρέπει να σα πω ότι χαιρετίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα θέλαμε αυτή η πρόταση να δοκιμήσει να αλλάξει το κείμενο της Κομισιόν όσο γίνεται λιγότερο. Να υπάρχει μια επιστηστική πτυχή στο πρόγραμμα και να βοηθήσουμε τους φτωχούς, τους ανήλικους, τους άστεγους. Τελικά έχουμε τον ελάχιστο κοινό παρομαστή των προτάσεων και γι' αυτό ευχόμαστε να μην αδυνατήσει πολύ η πρόταση Επιτροπής. Η προσέγγιση να κάνουμε αυτή τη κοινωνική πλαισίωση κατά του αποκλεισμού. Έχουμε κάποιε αλλαγέ στο κείμενο. Προτείνουμε κάποιε τροπολογίε. Ελπίζουμε ότι έτσι θα βελτιωθεί το πρόγραμμα. Και έχουμε συνεργαστεί για αυτό το λόγο με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η φτώχεια και η πείνα υπάρχουν παντού, σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα για τι πιο πλούσιε χώρε. Και η αλήθεια είναι ότι στι περισσότερε χώρε αυτή η πραγματικότητα γίνεται εντονότερη. Αυτό που θα συμφωνηθεί θα είναι αρμοδιότητα εθνική. Αλλά από πλευράς δαπανών θα φανεί τι κάνει κάθε χώρα, ποιες είναι οι αιτίε του φαινομένου, πώς θα πάει η Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι να, να γίνει κοινή εμπειρία το τι θα απογίνει το πρόγραμμα, κοινή εμπειρία που να αποκομιστεί από όλους. Είναι δείγμα αλληλεγγύης. Τα ευρωπαϊκά δεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι είναι μια πραγματικότητα. Ποια άλλο είναι και περισσότερο η φτώχεια και η πείνα. Θα στείλουμε επομένω ένα μήνυμα ότι τουλάχιστον κάπως έχουμε επίγνωση του τι γίνεται εδώ στα ευρώ τα γιατί αν δεν περάσει αυτή η πρόταση τότε το, το, το, το, μήνυμα θα είναι το μήνυμα της απομόνωσης, της αποξένωσης, τη αποστασιοποίηση. Κάτι άλλο θα σα πω αφορά το θέμα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, της φιλανθρωπίας κλπ. Γιατί ξέρουμε σε κάποιες χώρες που θεωρούν ότι αυτό είναι ισογύρισμα όσον αφορά την Ευρώπη, η οποία θα δίνει δέματα με φαγητά. Εντάξει, αυτό φαίνεται κάπως απλοϊκό, αλλά ο κόσμο θα πεινάσει να το κάνουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εκτό προγράμματο γίνεται σημαντικό έργο, όπω υπόθηκε πριν. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα τονώσει την αξιοπρέπεια του κόσμου. Ή το αντίθετο. Και αυτό ισχύει και για κάθε πρόγραμμα τέτοιο κοινωνικής αλλαγη Άρα, αυτή είναι η προσοχή που να κάνουμε. Κατά το αποκλεισμό, συμπερίληψη, κοινωνική λοιπόν πλαισίωση και να συνδυαστεί αυτό με άλλες πολιτικές. Και άρα με αυτό το πρόγραμμα να βοηθήσουν αυτούς που είναι περιθωριοποιημένοι να ενταχθούν και σε άλλα προγράμματα όπως και το πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου. πάση περιπτώσει, το εν λόγω, το συζητούμενο πρόγραμμα θα καλύψει πράγματα που δεν τα καλύπτει το ΕΚΤ. Έχουμε 14 τροπολογίες. Τώρα στο πεντέλεπτο που έχω δεν μπορώ να σας τα πω. Αλλά θα τις μοιράσουμε σε όλους. Θέλουμε να γίνει το κείμενο σαφέστερο, πιο αποδοτικό και θέλουμε την προσέγγιση του τύπου εταιρικής σχέσης. Να βαδίσουμε με αυτή την αρχή. Και έτσι να ευδοκιμήσει το πρόγραμμα Τώρα για τα τελευταία διαφορά που έχουμε, θα ήθελα απλώ να παίρνω μια το κοινοβούλιο ότι θα πρέπει το κοινοβούλιο να συνεχίσει να έχει την δυναμική του θέση. Και επίση πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να απευθυνθώ στου Γερμανού βουλευτέ και του Άγγλου, διότι η πραγματικότητα είναι ότι αυτή είναι η πλειοψηφία και οι χώρε σα ε, μετά να, να, να αναλάβουν και μπορούν να το κάνουν το πρόγραμμα. Να μην είναι οι χώρε σα στο, Συμβούλιο η παρεμπούδουσα μειοψηφία. Έτσι θα μάθετε πραγματικά. Μόνο με το πρόγραμμα αυτό τι γίνεται στην Ευρώπη. Αν δεν περάσει το πρόγραμμα θα είναι απίστευτα αρνητικό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπάλας Τσε, πρόεδρο της ε, Ένωσης για την Επιστημιστική Τράπεζα της Ουγγαρίας. Έχει το λόγο. Thank you. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι και εγώ μέλος ε, της ε, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τραπεζών τροφίμων και θα μιλήσω κατόπιν τούτου όχι μόνο για την Τράπεζα της Ουγγαρίας αλλά γενικότερα για το ευρωπαϊκό αυτό δίκτυο. Γιατί πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι σημαντικό, γιατί έχουμε 247 τέτοιες ε, τράπεζες ε, σε 21 χώρες και το 2011 διανύμαμε ε, σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη περίπου 429.000 τόνους τροφίμων. Το πρόγραμμα MDP για μας είναι ε, πάνω από το ίμιση των πόρων μας που είναι πολύ σημαντικό και η διανομή γίνεται με 31.000 ε, ε, φιλανθρωπικούς οργανισμούς και δήμους και κοινότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ανθρωπιστική, μάλλον με η ψητιστική βοήθεια είναι πολλαπλασιαστή. Αυτό αφορά ανθρώπου που έχουν ανάγκη, κυρίως το χειμώνα. Στην Ουγγαρία, παραδείγματο χάρη, οι τοπικοί δήμαρχοι μερικές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν φαγητό γιατί είναι αναγκασμένοι ε, να κάνουν αποταμιεύση και να ζεσταίνουν και τα σπίτια τους. Ε, εμείς λοιπόν είμαστε οι μόνοι μας λένε στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν. Όμως το πνεύμα της αλληλεγγύης στο οποίο αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό. Στο δικό μας το δίκτυο έχουμε όπως σας είπα 31.000 οργανώσεις και εκατοντάδες κοινωνικών λειτουργών χρησιμοποιούν την ε, βοήθεια με τρόφιμα για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν ανθρώπους μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει ένας κατάλογος προτάσεων που αφορά ε, στην αλλαγή, την τροποποίηση της πρότασης. Θα ήθελα να επισημάνω κάποια θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η μείωση του όγκου. Γνωρίζουμε ότι προβλέπονται περικοπές ε, του προπολογισμού από 3,5 δις σε 2,5 δις ευρώ. Όμως επιπρόσθετα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε μείωση του προϋπολογισμού. Ε, έρχονται νέες χώρες που προσχωρούν στο πρόγραμμα και με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ο αριθμός των χωρών που έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμά μας. Έτσι λοιπόν θα έχουμε συνολικά μια σημαντική μείωση ε, τροφίμων που διανέμουμε σε άτομα που έχουν ανάγκη. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώς μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε πια. Αυτό τώρα συζητάμε στην Τράπεζα Τροφίμων, ε, να δούμε ε, τι θα κάνουμε όταν θα υπάρξει σημαντική μείωση τροφίμων. Πώς θα μπορέσουμε να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν μπορούμε πια να σας βοηθήσουμε ακόμα και ε, μην ξεχνώντας ότι έχουμε και άλλους ανθρώπους που περιμένουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Ένα άλλο θέμα είναι η συγχρηματοδότηση που πρέπει να αποφευθεί. Υπάρχει, καταβάλλονται ήδη προσπάθειες στο πλαίσιο του προγράμματος. Το παλαιότερο πρόγραμμα ε, καλύπτει διοικητικής επίσεως θέματα και επιμελητίας. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του προγράμματος. Ε, αν δηλαδή ε, θέλει κανείς να μετακινήσει τα τρόφιμα, να τα διανύμει. Αυτό περιλαμβάνει συγχρηματοδότηση από εθνικές αρχές, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, την τοπική αυτοδίκηση και πάρα πολλούς οθελοντές. Υπάρχουν και όρια στο πρόγραμμα. Ορισμένες ε, οργανώσεις ε, έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα ή αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα λόγω του ότι υπάρχουν και όρια στη χρηματοδότηση. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι λάθος να υπάρχει επιπρόσθετη συγχρηματοδότηση. Ορισμένες χώρες ε, τελικά ίσως αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα και μάλιστα εκείνες που έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Ε, εμείς ε, διανέμουμε την βοήθεια σε τρόφιμα και ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικά χωριά όπου δεν έχουν τη δυνατότητα να δαπανίσουν χρήματα για την υποδομή. Εμείς λοιπόν ε, τους βοηθάμε να μοιράσουν τα τρόφιμα, πόσο μάλλον τώρα δεν θα ήταν παράλληλο να τους ζητήσουμε χρήματα στα πλαίσια της ε, συγχρηματοδότησης. Τώρα, ε, η, τα πλεονάσματα, κατά την άποψή μας, αυτό είναι ένα καθαρά οικονομικό θέμα. Πρέπει να δορίζεται αντί να καταστρέφεται, αλλά δεν πρέπει να αναμειγνύουμε αυτό με το θέμα της βοήθειας. Ίσως η λύση να είναι να υπάρξει διασύνδεση με το πρόγραμμα τροφίμων και οποροκυπευτικών που λειτουργεί σε κάποιες χώρες. Εάν υπάρχουν ε, ε, ε, ποσότητες στην παρέμβαση, αυτές μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν. Και το τελευταίο, η τελευταία διαφάνεια είναι εμείς πιστεύουμε ότι ε, το να επιληθούν τα προβλήματα και να ληφθούν αποφάσεις αυτό θα πρέπει να γίνει ταχύτερα. Το 2014 είναι πολύ κοντά, υπολείπονται πάρα πολλά για την προετοιμασία ενός νέου προγράμματος και εμείς θέλουμε διακαώς να συμπεριληφθούν και οι ΜΚΟ έτσι ώστε όχι μόνο η θεσμική αλλά και η επιτόπια γνώση να συμπεριληφθεί στο λειτουργικό σκέλος των μελλοντικών προγραμμάτων. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα, Γενική Γραμματέας της Eurochild, η κυρία Hainsworth. Ευχαριστώ. Είμαι η Τζάνα Hainsworth, Γενική Γραμματέας της Eurochild, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκό Οργανισμός, ε, ομαδικός που εκπροσωπεί ενώσεις και οργανώσεις που εργάζονται για τα παιδιά και τους νέους. Κατά πρώτον, ο Eurochild και τα μέλη, τα μέλη του δεν έχουν άμεση συμμετοχή από τα κράτη-μέλη Σημαντικό είναι ότι είμαστε και εμείς μέλος του MPM και συμφωνούμε με όσα είπε ο Φίνταν για το δικό τους δίκτυο. Θα ήθελα να σταθώ στα συγκεκριμένα σχόλια που έχω για το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο γενικές παρατηρήσεις δηλαδή. Πρώτα απ' όλα πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν θα αντιμετωπίσει το, πρόγραμμα, το πρόβλημα της ε, έλλειψης τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι σαν μια σταγόνα στον ωκεανό. Τα ποσά που προτείνονται είναι πάρα πολύ μικρά ω προ τι πραγματικέ ανάγκε που υπάρχουν. Στην Eurochild βλέπουμε να υπάρχει ένα όλο ένα μεγαλύτερο αριθμό παιδιών που δεν έχουν να φάνε, δεν μπορούν να πάνε σχολείο, δεν έχουν παπούτσια για να πάνε στο σχολείο, δεν έχουν θέρμανση. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υλική, υλικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Δεν θα αντιμετωπιστεί λοιπόν με το πρόγραμμα αυτό το φαινόμενο. Το άλλο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι ακόμη και αν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη υλικών πόρων, αυτό δεν θα άλλαζε κάτι ως προς την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Χρειαζόμαστε μια σφαιρικότερη, συνολικότερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της φτώχειας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά εντός αυτού του πραγματικού σκηνικού, τοπίου. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ευθεώς, διότι Εάν τα κονδύλια χρησιμοποιηθούν με τρόπο αποτελεσματικό, θα μπορούσαν να έχουν καταλητική επιρροή σε εθνικό επίπεδο και στο πώς σχεδιάζονται τα εθνικά μέτρα. Καταρχάς, να καλωσορίσουμε την προσέγγιση να περάσουμε από την επισητιστική βοήθεια σε κάτι πιο ευρύ, τα υλικά και μόνιμα αγαθά. Αυτό είναι μια πραγματική ουσιαστική διεύρυνση του προγράμματος Επίσης, η ηλική στέρηση για τα παιδιά είναι ένα θέμα που δεν θα μας απασχολήσει μόνο σήμερα, αλλά είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα για την κοινωνία μας και την οικονομία μας. Για τη διεύρυνση των προτεραιοτήτων του προγράμματος αυτό μας απασχολεί κάπως, διότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το πρόγραμμα είναι τόσο, ε, είναι τόσο, αποτελε... όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο επίση. Καλωσορίζουμε το συσχετισμό οποιασδήποτε παρέμβαση με την γενικότερη κοινωνική ένταξη των πλέον ενεκτούντων. Νομίζουμε ότι η διατύπωση τη πρόταση όπω αυτό είναι εύστοχη και χρειαζόμαστε ένα σαφή συσχετισμό με την, Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Ελπίζουμε ότι τις προσεχείς εβδομάδες θα έχουμε συγκεκριμένη σύσταση για την ε, παιδική φτώχεια και ευημερία, ε, όπως θα την καταρτήσουν και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Εδώ για τους δείκτες στην στέρηση υλικών αγαθών πρέπει να Είμαστε προσεκτικοί στον προσδιορισμό τους, ώστε το πρόγραμμα να χρησιμοποιείται και για αμοιβαία γνώση για να ανταλλαχθούν απόψεις και να δούμε γιατί η φτώχεια ως φαινόμενο διωγγώνεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φρικ. Σπίνεουάιν. Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με και για τους αστέγους. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Φρικ Σπίνεουεν και εργάζομαι για την Φιάντσα. Ε, uh, μια ομαδική, ένα ομαδικό οργανισμό που καλύπτει όσε ενώσει και οργανισμού εργάζονται για του αστέγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την Επιτροπή σα που μα έδωσε χρόνο ομιλία σε αυτή την τόσο σημαντική ακρόαση. Ωστόσο, νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν να έχουμε εκπροσώπου και από κάποιε από τι μεγαλύτερε οργανώσει που αυτή τη στιγμή εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματο, όπω τη Red Cross Caritas ε, Europa, δηλαδή τον Ερυθρό Σταυρό Κάριτα της Ευρώπης και άλλες οργανώσεις με σημαντικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα κάποια γενικά σχόλια. Καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα τη στηρίξει και θα παραμείνει κοντά στην αρχική πρόταση. Καλωσορίζουμε την έμφαση που δίνεται στην ακραία φτώχεια και τους πλέον ευάλωτους και την κάλυψη των ιατρικών τους αναγκών. Εδώ η διεύρυνση του πεδίου είναι σημαντική για να υπάρξει και ηλική στήριξη προς τους αστέγους, αλλά και τα παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Νομίζω ότι η έμφαση στους αστέγους είναι κάτι το υποχρεωτικό, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και την ε, παιδική φτώχεια. Η στέρηση επισητιστική είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα κάτι μέλη. Δεν γνωρίζω κανένα να γλιτώνει, κανένα τα κάτι μέλη να είναι απελαγμένο από αυτό είδου προβλήματα. Αυτέ είναι και συνέπειε τη κρίση βέβαια, αλλά και αναποτελεσματικών πολιτικών. Μην τα βάλουμε όλα στο ίδιο καλάτσι. Η κρίση είναι οξύτατη σε κάποιε χώρε. Σε κάποιες χώρες. 25% αυξάνονται τα ποσοστά των αστέγων σε χώρε όπω η Ελλάδα. Και βεβαίω αυτό συμπίπτει και με την πρόσφατη έμφαση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανεργία και την, ε, τον αποκλεισμό των νέων. Έτσι λοιπόν η ηλική στήριξη έχει επικεντρωθεί ως ένας ε, στόχος για την αντιμετώπιση της καταπολέμησης της φτώχειας ε, τα τελευταία 10 χρόνια και έχει συμπεριληφθεί και στην εμβληματική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της φτώχειας. Θα θέλαμε να παραμείνουν ε, οι στόχοι του προγράμματος κοντά σε ρεαλιστικά σκοπούς. Η πρόταση του προπολογισμού του προγράμματος είναι 2,5 δις. Ίσως να αυξηθεί εάν διαιρεθεί ο προτινόμενος προϋπολογισμός αν διαιρεθεί ο προπολογισμό που τώρα προτείνεται διά τον αριθμό των αστέγων που πραγματικά έχουν ανάγκη από στήριξη, θα φτάσουμε στα 3 ευρώ ετησίω. Χρειάζεται πραγματικά πολύ περισσότερα από το Ταμείο και θα πρέπει να προσέξουμε να μην παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό στο βασικό εργαλείο για να φτάσει η Ευρώπη του στόχου του 2020, δηλαδή να βγουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι από συνθήκε φτώχεια. Το Ταμείο αυτό το ESF και το ERDF δίνουν δυνατότητες στα κράτη-μέλη να διοργανώσουν περισσότερο δομημένε παρεμβάσει κατά τι φτώχεια. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εκμεταλλευτούν αυτέ τι ευκαιρίε. Εάν εντείνουμε τι φιλοδοξίε του προγράμματο αυτού, βέβαια, μπορεί να πληγούν οι πλέον ε, ευάλωτοι και οι πλέον μειονεκτούντε, που είναι και η ομάδα στόχο του προγράμματος. Έχουμε πάντως λόγους να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι σε επίπεδο Συμβουλίου θα υπάρξει επαρκής στήριξη για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε δεν θα μπλοκαριστεί, ελπίζουμε και θέλουμε να δούμε και δραστικές, να μην, δεν θέλουμε να δούμε δραστικές αλλαγές ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωκοινοβούλιο, διότι ήδη η ισορροπία στο Συμβούλιο είναι πολύ ευαίσθητη, έφραστη. Θέλουμε βεβαίως να γίνει δημοκρατική δουλειά όπως προβλέπετε, αλλά να έχετε υπόψη σε αυτή την περίπλοκη κατάσταση, γιατί ότι η συζήτηση για το Ταμείο να μην χρησιμοποιηθεί για την προσωπική προβολή κάποιων, αλλά για την κοινωνική πραγματικά ε, ωφέλεια που θέλουμε να προσφέρουμε. Επίση, υπάρχουν κάποιες βασικές, κάποιοι βασικοί περιορισμοί που που μας ε, αναγκάζουν να επικεντρωθούμε συγκεκριμένα στη σημεία του προγράμματο. Να αποφύγουμε τι επαναλήψεις και την επικάλυψη με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Να δούμε ε, την προστιθέμενη αξία του προγράμματο, του δημοσιονομικού περιορισμού, την ε, επιρροή που θα έχει στον τελικό καταναλωτή και ω προ όλου αυτού του περιορισμού να πω ότι θεωρούμε ότι η πρόταση τη Επιτροπή είναι και εύστοχη και επικαιρή παρά τη μείωση του προπολογισμού και προβλέπει την απαραίτητη διεύρυνση του πεδίου χωρί να υπερφορτώνεται το πρόγραμμα όπω προτείνεται. Νομίζουμε ότι η πρωτοβουλία εταιρική σχέση μπορεί να βελτιωθεί στην πρόταση, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλου εταίρου, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σκοπό είναι να αποτεχθεί και η άσκοπη γραφειοκρατία, που επίση είναι και τα πανηρή. Τέλο. Νομίζουμε ότι η καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απευθυνθεί προ τα κατεμέλη για το πώ θα χρησιμοποιήσουν σωστά το Ταμείο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα. Βάσει και των ε, γνώσεων των εμπειρογνωμόνων και των επιστημόνων, ώστε να ξέρουμε πώ να αναχαιτήσουμε τη φτώχεια, το πρόβλημα των αστέγων, την παιδική φτώχεια και την ε, έλλειψη επιστημιστική ασφάλεια. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε του πέντε εμπειρογνώμονέ μα. Είπα προηγουμένω πριν τι παρεμβάσει σα, ότι η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόληση δεν θα περιμένει την ψήφιση της έκθεσης της κυρία Κοστέλο για να δει αν θα υπάρξει πλειοψηφία υπέρ της ουσία της πρότασης. Διότι τώρα μιλάμε για την ουσία του Ταμείου. Αλλά υπάρχουν και όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε. Στη δική μας λοιπόν την ε, προσπάθεια Υπάρχει μια πραγματική δυσκολία. Μέχρι πού μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας και να παραμείνουμε στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή να συνεχίσει να ισχύει το γνωστό πρόγραμμα όπως ίσχυε και πριν, ή το κατά πόσον θέλουμε να μεταβάλουμε την προτινόμενη... το πρόγραμμα όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτάπητος, αυτό που εξετάζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Το λέω αυτό, γιατί όταν προτείνεται η πρικοδότηση του Ταμείου να μην συμπεριλαμβάνεται στην προκοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το, σημείο αυτό πιστεύω ότι χωράει πολλή συζήτηση. Βέβαια, είμαι πεπισμένη ότι ο προπολογισμό που προβλέπεται για το Ταμείο πρέπει να αυξηθεί. Διότι δεν ξέρετε κατά πόσον μπορεί να είναι ρεαλιστική άλλη πρόταση για χρηματοδότηση από την κοινή εγωτική πολιτική. Εδώ λοιπόν θα υπάρξουν ε, περίπλοκες και ενδιαφέρουσες διαπραγματεύσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Για την ώρα κανείς δεν έχει εγγραφεί στο κατάλογο των αγορητών. Βλέπω όμως τον κύριο Ορί και τον κύριο Σέρκας. Ήδη αρχίζουν να σηκώνονται χέρια. Κύριε Όρη. Σας ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε εδώ και κάνατε τις εγγύσεις σας. Δεν κατάλαβα καλά. Διατηρείται ακόμα και έπεισε επιφυλάξεις. Πώς θα εξεύρουμε μια λύση. Μια λύση που θα προβλέπει κάποια χρηματοδότηση. Ολική, μερικοί από πλευρά του Κοινωνικού Ταμείου. Εκεί έχετε δίκιο να έχετε τέτοιε επιφυλάξει γιατί φοβόμαστε. Και το έχουμε ξαναπεί. φορέ δώσει αυτά τα οποία δικαιούμαστε από το Κοινωνικό Ταμείο και ακόμα χρειάζονται χρήματα, οπότε θα πρέπει αυτοί οι οποίοι επιτόπου ασχολούνται με αυτή την υπόθεση είναι να, να μας πούν τη γνώμη του και να δούμε κατά πόσον αυτή η χρηματοδότηση ε, δεν θα έχει την τύχη που είχε στο παρελθόν. Τώρα, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τα θέματα που έχουν ε, σχέση με τη Γεωργία, την σχετική ε, αυτήν ε, επέμβαση τι θα γίνει με την ενσυπηστική βοήθεια ω προ την Γεωργία. Ε, ξεκαθαρίσουμε αν μπορείτε. Πώς η Γεωργία θα μπορούσε να συμβάλλει δηλαδή στην εμπιστική βοήθεια. Και αν υπάρχει σύγχυση μεταξύ διανομής ε, προκυπευτικών και εμπιστικής βοήθειας προς τους πλέον μειονεκτούντες άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Και πάλι χίλια ευχαριστώ για όλους όσους μίλησαν. Ε, Τώρα, οι βουλευτές, οι συνάδελφοι, αν θέλουν μπορούν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους πέντε εισηγητές μας. Όχι μόνο για τις απόψεις τους, αλλά και για το έργο το οποίο επιτελούν. Παντού, σε όλη την Ευρώπη. Η ανθρωπιά λείπει στις μέρες μας, οπότε έχει ακόμα μεγαλύτερη αυτό το οποίο κάνουν. Αυτά χρειάζονται την ώρα της κρίσης. Μια που έχει γίνει δυσδιάκριτη ε, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανθρωπιζ... ανθρωπιάς και, και, και βαρβαρότητας. Μας είπαν την ανησυχία τους. Συμφωνώ μαζί τους. Ότι το τοπίο είναι γεμάτο με ερωτηματικά. Τι θα γίνει με το Κοινωνικό Ταμείο. Στο μέλλον θα είμαστε δίπλα σας εμείς σοσιαλιστές, αλλά να μην ξεχνούμε, να μην ξεχνούμε, να μην παραλείπουμε, να λάβουμε υπόψη ότι όσες δυσκολίες είναι τόσα χρόνια, γιατί υπάρχει τόσος κόσμος που θέλει ε, ε, προθύμως να καταστρέψει την ε, Ευρώπη. Και το κάθε κράτος να πορεύεται μόνο του. Εντάξει, έχουμε αφετηρία τώρα από τη Επιτροπή. να δούμε όλες τις αναλεκτικές, όλες τις δυνατότητες επί τη βάση αυτής της πρότασης της Κομισιόν. Είμαστε ρεαλιστές, το ξέρετε κι εσείς όπως το ξέρουμε και εμείς και στο καλύτερο από εμάς, ότι αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι πολύ πιο αξιόλογο από ότι κάθε θεωρητικολογία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ομιλητές. Ε, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λιγάκι και έχασα την πρώτη ομιλία. Αλλά είχα ήδη μιλήσει στους ε, συναντέλφους σας. Ε, συναντήθηκα μαζί τους πριν από δύο εβδομάδες. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά τη δουλειά που κάνετε. Κάποια σχόλια και κάνα δύο ερωτήσει θα κάνω. μιλήσατε για την αξιοπρέπεια και φαντάζομαι και για την αυτονομία του ατόμου, το πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Επίσης, η κυρία Hensworth μίλησε για ένα μικρό ποσό χρημάτων ε, που ε, χρησιμοποιείται σωστά. Ή δυνατόν, θα ήθελα λιγάκι να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς εννοείτε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά θα ήθελα όλα αυτά να τα συνδυάσετε με το ταμείο για το οποίο συζητάμε σήμερα εδώ. Επίσης, ε, ε, ο τελευταίος ομιλητής ε, μίλησε για την καθοδήγηση που πρέπει να υπάρξει σχετικά με το Ταμείο. Τα σχόλιά μου είναι τα εξή. Πρέπει να δείξουμε στους Ευρωπαίους ότι υπάρχει προστέμενη αξία. Εχθέ διάβασα λίγο τι τελευταίες γνωμοδοτήσεις από την, τη Βουλή της Αγγλίας το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Και ε, σκέφτηκα λοιπόν η στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και η στόχοι για τη μείωση της φτώχειας. Αν διαβάσετε αυτές τις νομοθετήσεις, ε, κυρίως ε, τη, της Βουλής Αγγλίας, της Κατοβουλής, ε, θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότεροι από εμά, όχι όλοι, αλλά πιστεύω οι περισσότεροι, στηρίζουν αυτό το ταμείο. Και άκουσα αυτά που είπατε για την μειονότητα που μπλοκάρει. Ε, Πρέπει λοιπόν επιχειρήματα να προβάλλονται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Ο συνάδελφος από την Ουγγαρία μας είπε ότι οι άνθρωποι δεν περισσεύουν λεφτά να φάνε γιατί πρέπει να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Ε, θεωρώ ότι όλα αυτά που λέξανε είναι πολύ σημαντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ίσως μπορείτε αυτά που μας είπατε να τα συσχετίσετε με κάτι το πιο συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κορνέλισεν, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές ε, για τις πληροφορίες που μας ε, έδωσαν. Ε, πραγματικά συμφωνώ με όλους αυτούς που πιστεύουν ότι θα πρέπει να λάβουμε περισσότερα διαρθρωτικά μέτρα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζουν με λιγότερη φτώχεια. Βέβαια, από τη μια πλευρά πολλές οικονομικές πολιτικές οδηγούν τους ανθρώπους όλο και περισσότερο στη φτώχεια. Ε, και τώρα τι κάνουμε, ε, φτιάχνουμε ένα μικρό ταμείο για να προσφέρουμε κάποια τρόφιμα. Αλλά όμως ε, δεν λαμβάνουμε τα απαραίτητα κοινωνικά μέτρα που θα έπρεπε να λάβουμε. Πάντως η κατάσταση αυτή τη στιγμή αυτή είναι και κατά τη δική μου άποψη το σημαντικότερο όλων είναι να διασφαλίσουμε ότι το ε, Ταμείο δεν θα πάψει να λειτουργεί απότομα την 1η Ιανουαρίου του 2014. Κατά την άποψή μου αυτό σημαίνει ότι ε, πρέπει να ε, τροποποιήσουμε το Ταμείο εκβάθρων για να βρούμε μια λύση και με το Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ταμείο. Το Συμβούλιο είναι αντίθετο και υπάρχει μια μειονότητα που μπλοκάρει. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι αυτή, αλλά φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε λιγάκι το πώς κατανέμονται τα κονδύλια. Ε, όπως ανέφεραν κάποιοι ομιλητές, ε, αν όλες οι χώρες αρχίσουν να συμμετέχουν, τότε δεν θα απομένουν και πάρα πολλά για τις ε, τράπεζες ε, τροφίμων, από τις οποίες τώρα εξαρτώνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε το Ταμείο ε, και ίσως κύριε Φορέλ, ίσως μπορείτε να μας απαντήσετε τι πιστεύετε. Δηλαδή, θεωρείται ως ε, βάση ε, για ε, την περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων θα χρησιμοποιήσετε μόνο την κοινωνική ένταξη. Κοιτάξτε, όταν είναι κανείς άνεργος δεν ξέρω αν υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο. Το δεύτερο που πρέπει να εξετάσουμε είναι η επικουρικότητα. Άκουσα από τον συνάδελφό μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο στην Ολλανδία ότι υπάρχει μια συζήτηση για αυτό το ταμείο ακριβώ τώρα που συζητάμε και εμείς. Και εκεί ο η Υφυπουργό είπε ότι ε, μπορεί να ε, σκεφτεί το να γίνει πιο επικοδομητική, να εγκαταλείψει την μειονότητα που μπλεκάρει, εάν πρόκειται για ένα ταμείο μεταβατικό, όπου οι χώρες ε, που το χρησιμοποιούν τώρα θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν και μετά από 7 χρόνια το ταμείο ε, να συρρυκνωθεί. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι θα υπάρξει και χρόνος για να γίνει το ταμείο ανεξάρτητο. Ε, απευθύνομαι στον Ούγκρο συνάδελφο. Από αυτά που μας είπατε, ε, φαντάζομαι ότι θέλετε να υπάρχει αυτό το ταμείο για πάντα. Ε, τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να προσφέρουμε από πλευράς ε, εγκαταστάσεων ε, και υποδομής ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τι μπορούμε να προσφέρουμε έτσι ώστε να μπορείτε μετά από 7 χρόνια να είσαστε ανεξάρτητοι από την επισητιστική βοήθεια. Και για να βοηθήσω λιγάκι και τη συζήτηση, θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει τελικά εάν το Συμβούλιο μπλοκάρει και το ε, Ταμείο πάψει, πάψει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου του 2014. Καρή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία κυρία Κυρία Πρώτα πρώτα. Να ευχαριστήσω όλους τους φορείς για τόσο να μας είπαν, αλλά κυρίως να τους ευχαριστήσω για την κινητοποίηση. Αυτό που κάνουν για να σώσουν ό,τι μπορεί να σώθει. Να έχουμε δηλαδή ένα τέτοιο καινούργιο ταμείο για την εμπιστική βοήθεια. Χωρίς να κινητοποιηθεί ο κόσμος, νομίζω ότι ακόμα. Και έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε. Ακόμα και αν η Επιτροπή μας τάξει ως προτεραιότητα αυτόν τον αγώνα κατά της πείνας κλπ. Ακόμα και αν έχουμε αυτή εδώ την πλατφόρμα της, της πάλης, χωρίς Χωρί λοιπόν να δεν γίνει κάτι άλλο. Αν δεν καταλάβουν τα κράτη ότι χρειάζεται κάποια στρατηγική, δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να γίνει αυτό προτεραιότητα. Και εγώ λοιπόν χαιρετίζω και, και νιώθω ανακούφιση το ότι προτείνεται αυτό το νέο ταμείο. Χρειάζεται αυτή η βοήθεια και όπως είπε η συνάδελφο, δεν ναι, αρκεί αυτό γιατί σήμερα δεν χτυπάμε άμεσα και τις ρίζες του κακού, της φτώχειας. Και ακριβώς όπως είπαμε για αυτή την πλατφόρμα της καταπολέμησης της φτώχειας ε, και αυτή τη στρατηγική 2020 σημαίνει ότι πρέπει να, να, να, μειώσουμε αυτούς τα, 20 εκατομμύρια τους, τους φτωχούς με το 2020. Άρα χρειάζονται εργαλεία, μέσα, ε, ελάχιστο εισόδημα κλπ. Άλλο θέμα αυτό. Τώρα όσον αφορά το Ταμείο. Βεβαίως Νομίζω ότι η επέκταση, η παρέκταση τέλος πάντων του, του, του, του, του ε, της δράσης είναι σωστή και εγώ ε, χαιρετίζω το ότι δίνουν προτεραιότητα στους αστέγους. Γιατί, γιατί εγώ, ξέρετε, ε, ε είχα ξεκινήσει αυτή την, την, ιδέα για τους αστέγους, αλλά όμως ε, όπως είπαμε πριν αυτό είναι μία μια σταγόνα το ωκεανό. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό το ταμείο θα πρέπει να συνοδευτεί, να, να, να πάνε, πάνω από δύο χρόνια που την, την ε, πολιορκούμε επί την Κομισιόν για να φτιάξει, να προτείνει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους ε, αστέγους και να υπάρχει ένας, ένας χάρτης πορείας για όλα τα κράτη. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα αν δεν υπάρχει μια στρατηγική. Τώρα όσον αφορά τα της εμπιστικής βοήθειας, αυτό φυσικά θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό είναι καθημερινή επίγουσα ανάγκη. Χρειάζεται μια τέτοια πολιτική επομένως η οποία θα σώσει ζωές και θα μην το ξεχνάμε. Και επίσης να σας πω ότι ε, όντω υπάρχει εδώ πέρα κάποια σχέση με την κοινή ε, γεωργική πολιτική, διότι σήμερα αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι δεν υπάρχει πλέον πλεόνασμα όσον αφορά τα, τα, τα τρόφιμα. Άρα θα πρέπει τα κρατημέλη να, να κάνουν αυτό που είναι ο ρόλος τους, δηλαδή να, να, να ασκήσουν την σωστή τιμολογική πολιτική. Και εμεί επίση θα πρέπει να πιέσουμε μέσω της Επιτροπής ε, γεωργία και έτσι να υπάρχει ένα μέσον, ε, να υπάρχει ε, κάποια νομοθεσία δηλαδή για να μην έχουμε εκτείναξη των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Πρόκειται όμως τώρα για μια ευκαιρία που έχουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε αποκεντρωμένα να τρέξουμε κάποια καινούργια προγράμματα. Ε, στη Γαλλία υπάρχουν περιφερειακά, καινοτόμα, οικολογικά, όπως το Πουατού Σαρόντ. Αυτό με αυτά τα προγράμματα συνδέονται οι τράπεζες οι διατροφικές, η τοπική γεωργία, υπάρχουν τα μπακάλια της ελληνικής και οι στόχοι είναι πολλαπλοί. Πρώτα-πρώτα έτσι οι πιο μειονεκτούντες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια υγιεινή διατροφή και με τακτική ε, διανομή ο επίσης. επίσης. Είναι πάρα πολύ μεγάλες και σοβαρές οι επιπτώσεις στην υγεία. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε. Να ενισχύσουμε τη σχέση παραγωγού καταναλωτού. Και έτσι θα αναδειχθεί και η τοπική γεωργία. Επομένως, με κάποια ρύθμιση, πρόβλεψη, νομοθεσία μπορούμε να έχουμε όντως κοινωνική ένταξη, κοινωνική πλαισίωση και έτσι με αυτή την το τοπική, την, την, τη γεωργία, την κοντινή όπως τη λέμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Θυμάμαι τι είπε ο κύριος Φάρελ πριν. Είπε προσοχή να μην γλιστρήσουμε σε μια συζήτηση για την φιλανθρωπία προσοχή, μην, ε, μην έχουμε εδώ πέρα ναρκοθέτηση και υπονόμευση. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή ελληνική που είναι κάτι πολύ πολύ ευρύτερο. Είναι το δικαίωμα του να ζει κανείς με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το χρειάζονται. Τώρα, πρόεδρε, το είπατε. Τι θα, μήπως χρειάζεται να έχουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο και όχι να εντάξουμε αυτή την ε, δράση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. το πρώτο θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει με τίποτα αυτό το καινούργιο ταμείο ε, να ε, το, έχουμε τόσο το έχουμε, το έχουμε κάνει τόσο τόσο ε, ανελαστικά φτιαγμένα να λέμε τόσο ποσοστό για άνεργους τόσο για άστεγους κλπ. Όχι. Να, υπάρχει, να υπάρχουν περιθώρια ελιγμών, να υπάρχει ευελιξία γιατί ας πούμε, μπορούμε να πούμε στη Γαλλία 15% θα δίνουμε στους άστεγους, ξέρω εγώ, 5% να, να λένε στην Ελλάδα. Πρόκειται για, για συγχρηματοδότηση. Έτσι κι μιλούμε για κλίμα ε, λιτότητας. Πρόκειται επομένω. Για, κάθε χώρα πρέπει να έχει τι δικέ προτεραιότητε και επομένω θα πρέπει η χρηματοδότηση να πηγαίνει στου διάφορου φορεί. Και αυτό σα το λέω, γιατί τώρα ο, ο μείζον κίνδυνο είναι οι διαπραγματεύσει. Οι διαπραγματεύσει, οι δημιουργικέ όσον αφορά την κάλυψη αυτού του, του ταμείο, γιατί εάν δεν συνεχίσει να υπάρχει το ταμείο ή τουλάχιστον να ακόμα περισσότερο, τότε τι θα κάνουμε. Και αυτό τώρα είναι ο κίνδυνο σήμερα, ότι θα πρέπει ε, ε, τώρα να, να, να προλάβουμε αυτέ τι εξελίξει. Κινητοποίηση. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο επομένω να τοποθετηθεί και να πιέσει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Σρέτερ. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη ερώτηση προς τους ε, εμπειρογνώμονες. Ε, αυτό το ταμείο μέχρι τώρα έχει ένα σταθερό ε, προϋπολογισμό. Δεν συμμετέχουν όμως εκεί όλα τα κράτη, απλά συμμετέχουν κάποια μέσα από την επισητιστική βοήθεια. Το νέο ταμείο ε, είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει πρόγραμμα σε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και σε πλούσια, όπως είναι η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία, που όμως ε, έχουν μια, έναν πολύ έντονο διαχωρισμό ανάμεσα στους ε, πλούσιους και τους φτωχούς. Κατά την μου λοιπόν αυτό ε, δεν είναι σωστό διότι το οικοδόμημα είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που κατ' ουσίαν σημαίνει ότι έχουμε μία ανακατανομή σε αυτό το ταμείο από εκείνες τις χώρες που μέχρι τώρα το χρησιμοποιούσαν και όπου εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από την ευρωπαϊκή βοήθεια, φεύγουμε από αυτό και πάμε σε εκείνες τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τοπικές πρωτοβουλίες, με τοπική χρηματοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση και ξαφνικά αρχίζουν να εμφανίζονται κοινοτικά κονδύλια. Εσείς τι πιστεύετε, πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί εγώ έχω ε, μεγάλες ε, επιφυλάξεις ως προς αυτό το ταμείο. Δηλαδή υπάρχει η κατάσταση όπου από το 20% που το αποκτήσαμε με κόπο να δαπανώνται χρήματα σε τομείς οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν εθνικά χρηματοδοτούμενοι και αυτά τα χρήματα απλά ε, θα αντικαταστήσουν τα εθνικά φιλανθρωπικά ειδήματα και την εθνική υποστήριξη. Ε, και οι χώρες που αναφέρονται στον πίνακα αυτές ε, κατ' ουσίαν θα λάβουν ε, μικρότερα κονδύλια, όχι διότι απαραίτητα το Ταμείο ε, θα έχει μικρότερη πρικοδότηση, αλλά διότι θα συμμετέχουν περισσότερες χώρες. Και υπολογίσαμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι η Γερμανία θα παίρνει 50 εκατομμύρια το χρόνο και η Μεγάλη Βρετανία μάλιστα 38. Άρα δηλαδή αυτό θα αφαιρεθεί από άλλες χώρες που οι άλλες χώρες έτσι και αλλιώ ε, στο μεσοπρόθεσμο ε, σχεδιασμό θα υποστούν περικοπές. Πρέπει να σας πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η απάντησή σας σε αυτά που σας ρώτησα. Η κυρία Μπάουα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση για τις επισητιστικές τράπεζες. Δεν είμαι μεν Δήμων, αλλά κατάφερα να διαβάσω κάποια πράγματα και να τα μελετήσω. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό πώς ε, θα ε, διαμορφωθεί, πώς θα σχεδιαστεί ώστε να περνάει η επιστημιστική βοήθεια εκεί που πρέπει, να φτάνει στο στόχο της. και επίσης για τις ενώσεις ε, του που θα πρέπει να υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν εθελοντές πώς θα λειτουργεί ακριβώς μια επισκεπτική τράπεζα Πρόεδρος, ευχαριστώ Κυρία Κοστέλο, θέλετε να θέσετε ερωτήσεις στους παρεμένοντες Θέλετε να ρωτήσετε κάτι Πρόεδρε, θα ήθελα μια ευκαιρία να συνοψίσω στο τέλος. Πριν την ανακεφαλαίωση, μήπως έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους παρεμβαίνοντες για τις παρουσιάσεις τους. Οι ερωτήσεις που έχω έχουν να κάνουν με, τη διαχει... με το πώς θα διαχειριστούμε την πρόταση ανυπομονούμε να δούμε και τις τροπολογίες που θα υποβληθούν, αλλά και τις δικές σας προτάσεις για να βελτιωθεί το πρόγραμμα να ενσωματώνονται. Ένας από, το στο... τους τομείς που όλοι θίξατε ήταν όσοι έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του προγράμματος. Ιδιαιτέρως, ήθελα να ξέρω ποιε είναι οι απόψεις σας για τη διαχείριση του προγράμματος όπως τώρα προτείνεται, σε σύγκριση με το τι ίσχυε προηγουμένως έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια απλούστευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πολλά από αυτά που προτείνονται θα καθησυχάσουν φόβους και ανησυχίες για περί το γραφειοκρατικό άχθος. Είχατε τη δυνατότητα να δείτε κατά πόσον αυτό ισχύει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης σημειώνω ότι ο καθένας από τους ομιλητές είπαν, είπε ότι ανησυχεί για τη συνέχιση του προγράμματος. Όπως είδατε και εμείς θέλουμε να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι η διεύρυνση του πεδίου του προγράμματος. Ασχολούνται και με νέα θέματα όπως η στέρηση υλικών αγαθών. Είπατε ότι Γενικώ σα ικανοποιούν οι τομεί που στοχεύονται. Ε, και τελικώ με τα μέτρα συγχρηματοδότηση. Οι στόχοι του προγράμματος για την στέρηση τροφίμων, την παιδική φτώχεια και του αστέγους είναι στοιχεία που πιστεύετε ότι καλύπτονται παρκώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ να ανακεφαλαιώσουμε τις ερωτήσει μας. Πιστεύω βέβαια ότι προσκεκλημένοι τι σημείωσαν. Εμένα με ανησυχεί το εξή βλέποντας με τι πίεση εκπώνησε το πρόγραμμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έλεγα ότι ο κίνδυνος είναι διτός. Πρώτον, να μπούμε σε μια λογική κονδυλίων εφόσον αρχίζουμε να μιλάμε για συγχρηματοδότηση. Δύσκολο θα είναι να επιτευθούν οι στόχοι των επισητιστικών τραπεζών. Οπότε, από εσάς ήθελα να μου πείτε, δεδομένων των νομοθετικών περιορισμών <clears throat> λόγω των νομοθετικών περιορισμών, ιδίω τη απόφαση του δικαστηρίου. Δεδομένου λοιπόν αυτού του εμποδίου, Πώ θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Δεύτερη ερώτηση. Η διεύρυνση του πεδίου με στόχους φτώχειας πλέον. Κατά της φτώχειας δηλαδή. Μήπως ε, αποδυναμώνεται η ουσία, ε, γίνεται πιο αδύναμη η δυνατότητα παρέμβασή σας. Θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο νομίζω. Θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συζητήσουμε την έκθεση της κυρίας Κοστέλλου. Νομίζω μπορείτε να απόσχετε για την ώρα. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στους ομιλητές μας για τις απαντήσεις τους. Βέβαια θα είναι δύσκολο γιατί ήταν πολύ άριθμες ερωτήσεις και δεν είναι πολύ ο χρόνος που θα σας δώσω. Πέντε λεπτά ο καθένας σας. Ας ξεκινήσουμε αντιστρόφως από ό,τι προηγουμένως. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Φρικ Σπίνεβαϊν. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με αστέγους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Το ερώτημα για το κατά πόσο το πρόγραμμα θα πρέπει να στοχεύει περισσότερο σε φτωχότερες χώρες από τις πλήσεις. Αυτό είναι πλούσιες, είναι δύσκολο να απαντηθεί. Βέβαια, ε, είπαν και άλλοι ομιλητές προηγουμένως ότι το θέμα της έλλειψης στέγης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αν τελικά στοχεύει κανείς ε, στους αστεγούς ε, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χρησιμοποιώντας διάφορες λύσεις, ίσως όχι απαραίτητα οικονομικές. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια ερώτηση παγίδα. Τώρα, όσον αφορά στη διεύρυνση του πεδίου. Είπα ήδη προηγουμένως ότι κατά την άποψή μας είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η διεύρυνση, έστω και σχετικά περιορισμένη, δηλαδή είναι απόλυτα σαφές ότι σε κάποιο βαθμό όλα αυτά θα γίνουν εις βάρος εκείνων που πήγαν προηγουμένως για την επιστημιστική βοήθεια. Νομίζω όμως ότι η διεύρυνση έχει ως στόχο και κάποια καλή βούληση από πλευράς κρατών μελών. Υπάρχουν στρατηγικοί λόγοι γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ε, διεύρυνση του πεδίου. Υπήρξαν πολλές ε, ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της πρότασης, κατά πόσον μπορούν να εφαρμοστούν μερικά πράγματα από νέους τομείς όπως είναι η παιδική φτώχεια και το πρόβλημα των αστέγων. Πρέπει να είμαστε όμως και επικοδομητικοί. Η δική μου οργάνωση ήδη προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα ε, να δημιουργηθούν πακέτα ε, αρχικά. Δηλαδή να βοηθάμε στην αρχή να τους βάζουμε σε ένα σπίτι και αυτοί όμως δεν έχουν τα βασικά για να επιβιώσουν. Δεν έχουν ας πούμε εργαλεία κουζινικής ή καθαριστικά ή έστω κάποια έπιπλα. Και σε πολύ λίγες χώρες ε, μπορεί κανείς, ε, υπάρχει δυνατότητα όλα αυτά ε, να μπουν σε ένα πακέτο και να προσφερθούν σε έναν άστεγο που μπαίνει σε ένα σπίτι. Εμείς κάναμε έναν υπολογισμό ε, πόσο κοστίζει αυτό γιατί βεβαίως ε, υπάρχουν διάφορες ε, προσφορές και τελικά αν μπει κανεί στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με 25 εκατομμύρια μπορεί κανείς να καλύψει αν θέλετε ένα μεγάλο κομμάτι των αστέγων που είναι σε αυτή τη μεταβατική φάση. Ε, βρίσκουν κάποια ε, στέγη και εκεί τους προσφέρει κανείς αυτό το ε, βασικό πακέτο για να επιβιώσουν. Με λίγα λοιπόν χρήματα μπορεί κανείς να επιτύχει κάτι σημαντικό σίγουρα στον τομέα των αστέγων. Άρα δηλαδή υπάρχει και δυνατότητα να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που προτείνουμε. Ευχαριστούμε κυρία Χένσουαρθ, για τον Eurochild. Σας ευχαριστώ. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Δεν θα απαντήσω αναγκαστικά στα, προγράμματα, στα προβλήματα για την διαχείριση του προγράμματος, αλλά για την διεύρυνση του προγράμματος και σε άλλους τομείς. Επειδή ξεφεύγει από την επιστημική βοήθεια πια. Η προτεραιότητα για να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια. Νομίζω ότι συνάδει με τι πολιτικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πολέμηση τη παιδική φτώχεια. Όπω είπα προηγουμένω, και λόγω τη άμεση ανάγκη των παιδιών, αλλά και λόγω τη ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό ο φαύλο κύκλο μειονεκτούντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιστιστική βοήθεια και το σχετικό πακέτο και το περιεχόμενο του προγράμματος αυτού, με αυτό το νέο στοιχείο, όντω θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια υγεία διατροφή και μακροπρόθεσμη ένταξη παιδιών και νέων. Έπειτα έγινε μια παρατήρηση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο αυτό με τρόπο ευφυή και πώς μπορεί να ενισχυθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να μην είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα δηλαδή, αλλά ένα χέρι βοηθείας. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή ε, γίνεται σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι συμπληρωματικό και πρέπει να ενισχύσει το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα των παιδιών και πρέπει να δοθεί έμφαση στην υλοποίησή του. Οι εμπλεκόμενοι να χρησιμοποιήσουν το ταμείο αυτό ως συνοδευτικό μέτρο να δώσει δηλαδή μακροπρόθεσμε λύσει για την διέξοδο από τι συνθήκε φτώχεια. Και έπειτα για τι δείκτε. Έγινε μια παρατήρηση για τη χρήση των δικτών για τα νοικοκυριά όπου και δύο είναι άνεργοι, για την ηλική στέρηση, για την ενεργεία των νοικοκυριών εδώ ε, καλώ συμπεριλήφθη αυτό ο στόχο του Ταμείου και επίση η στέρηση υλικών αγαθών αφορά ιδιαίτερα το, θέμα της, το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας όπως με το πρόγραμμα ΣΥΛ και τους δείκτες που πρόσφατα ε, είδαμε να δημοσιεύονται. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό θα πρέπει να συναποτελέσει μέρος των στόχων του προγράμματος. Ευχαριστώ. Κύριος Τσε, ευχαριστώ. Να προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω στην ερώτηση για το ποιο είναι ο ρόλος των επισητιστικών ε, τραπεζών και τη χρήση του προγράμματο. Οι επισητιστικέ τραπεζέ, μαζί με άλλε οργανώσει, ε, προσπαθούν να διοργανώσουν και να διαχειριστούν την διανομή τροφίμων καθώς και τη συλλογή τους. Υπάρχουν περίπου 500 τέτοιες οργανώσεις στην Ουγγαρία. Εκείνες, χάρη σε εμάς, λαμβάνουν τα τρόφιμα τα οποία μετά μπορούν να προωθήσουν στο κοινωνικό τους στο, σκέλος, στο κοινωνικό σκέλος του έργου τους. Είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συλλέγουμε τρόφιμα και τα διανέμουμε στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες επιλογές μας, τι άλλες δυνατότητες έχουμε δηλαδή εκτός του προγράμματος για να ενισχύσουμε τις επιστητικές τράπεζες, έχουμε και άλλες σημαντικές πηγές όπως τα πλεονάσματα της διατροφικής αλυσίδας, της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό διότι πραγματικά τα πλεονάσματα θα μπορούσαν εύκολα να μετατρέπονται σε επισητιστική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη νομίζω ότι σπαταλούμε εκατομμύρια τόνων τροφίμων. Αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτή είναι μία από τις αφέστερες αρμοδιότητες των επιστημιστικών ε, τραπεζών. Δηλαδή να εντοπίσει τα πλεονάσματα αυτά και να εξεύρει νέες πηγές ε, επιστημιστικής βοήθειας. Βέβαια, δυστυχώς εδώ έχουμε κατά προσέγγιση δεδομένα και όχι ακριβείς αριθμούς για τα πλεονάσματα, ώστε να δούμε τι δυναμικό θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε Ίσως να μπορούσαμε να βελτιώσουμε εδώ τους στόχους συνεργασίας της ε, βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων με τις δημόσιες αρχές και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που σε κοινωνικό επίπεδο παρεμβαίνουν στην όλη προσπάθεια. Υπάρχουν κάποια μικρότερη εμβέλειες προγράμματα στην Ευρώπη, τα οποία θα μπορούσαν να προβληθούν περισσότερο και να έχουν ε, επιπτώσεις ε, χιονοστιβάδας, να λειτουργήσουν δηλαδή σορευτικά. Πάντως, για την επιστηστική βοήθεια σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, οι δωρεές που προέρχονται από τα επιστηστικά πλεονάσματα ε, υπόκεινται σε ΦΠΑ. Φορολογούνται οι επιχειρήσεις, έχουν ε, περισσότερο όφελος οικονομικό εάν καταστρέψουν τρόφιμα παρά αν τα δωρήσουν. Αυτό ουσιαστικά δυσκολεύει τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που μπορούν να βελτιωθούν. Πέραν αυτού, είναι σημαντικό στοιχείο και η ευαισθητοποίηση. Θα θέλαμε ένα ευρωπαϊκό έτος ε, κατά της ε, κατασπατάλησης τροφίμων να προβλεφθεί και αυτό διότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με αυτήν την αφορμή προγράμματα ώστε να βρεθούν περισσότερες συμπληρωματικές πηγές τροφίμων πέραν του προγράμματος FIT και να ενισχύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Κύριος Φάρελ, υιοθετούμε τη σκοπιά... Όμως, άλλοι εμπλεκόμενοι και συνεργάτες μας κάνουν τη διαχείριση, έχουν συγκεκριμένες πληροφορίε. Αυτό το οποίο είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το συζητήσαμε και για τις ερωτήσεις σας έχουμε τις απαντήσεις. Σε πέντε λεπτά δεν γίνεται αυτό. Οπότε να πάτε να βρείτε παρακαλώ αυτές τις οργανώσεις. Αυτούς που ε, ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' για, για την πρικοδότηση. Εσείς εδώ στο Κοινοβουλίο, νομίζετε ότι μπορείτε να έχετε καλύτερη πρικοδότηση, τέλειο. Μπορείτε όμως να το κάνετε. Πολύ καλό. Τώρα όσον αφορά το Νομικό μέσο, ναι, το είναι σαφές τώρα, διασκεδάστηκαν οι αμφιβολίες, όμως θα πρέπει να γίνει πλαισιώση μέσω του ΕΚΤ, γιατί πρέπει όλος ο κόσμος να καλυφθεί και οι νέοι να έχουμε άμεσα την παροχή βοήθειας. Γίνεται αυτό με τον κανονισμό που διέπει το ΕΚΤ. Δεν νομίζω αυτό νομικά ότι γίνεται, γιατί είναι σαφή, σαφέστατη η νομική βάση εκεί πέρα. Οπότε, εάν τελικά δεν έχετε κάποιο συγκεκριμένο μέσο, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνει, καν, να μην τίποτα. Οπότε είχαμε αυτό το 12% του κοινωνικού ταμείου για την κοινωνική, τον κοινωνικό αποκλεισμό και όλα αυτά. Προσοχή εκεί, να μην ε, έχουμε από εκεί καταστροφή. Αυτό το 20% να είναι επιπλέον χρήματα. Είναι διαφορετικό το πρόγραμμα τώρα και νομίζω ότι γιατί πρέπει να είναι ξεχωριστό πρόγραμμα, είναι μια ξεκάθαρη νομική βάση. Κάτι άλλο επίσης όσον αφορά κάποια ευφυή χρήση αυτού του ταμείου. Πρώτα-πρώτα, πρόκειται τώρα για σημεία επαφή με αυτούς τους τόσο ευάλωτους. Να τους οδηγήσουμε και σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται. Αυτό λένε εννοούμε έξυπνη χρήση του Ταμείου. Άρα είναι σημείο επαφή πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Οι τράπεζες ε, συμπεριλαμβάνουν τον κόσμο σε αυτή την, την, την διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Πολλά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Αυτό εννοούμε επομένω σχεδιασμό και χρήση ευφύ. Τώρα, με αυτές τι αιτιολογημένες ε, γνώμες, στην Bundestag και στο House of Lords, τελικά ε, επικαλούνται την ε, επικουρικότητα. Το θέμα όμως δεν είναι το αν θα λύσουμε γενικά την πείνα, τη φτώχεια αυτά. Μιλάμε για μια συμβολή απλώς. Αλληλεγγύη στην προσέγγιση. Να μάθουμε Γι' αυτό είναι σημαντικό όλες οι, να εμπλέκονται οι χώρες. Ε, αυτό θα πρέπει να δούμε. Γιατί έχουμε το, το θέμα αυτό. Γιατί έχουμε την ανάγκη για χρήματα. Γιατί έχουμε την πείνα. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να αλλάξει το σύστημα, να έχει πιο συστημική προσέγγιση και όλες οι χώρες να δουν κατά, κατά πρόσωπα την, την, την πραγματικότητα. Επομένω, ο ένα να διδάξει στον άλλο ποιοι είναι οι πιο έξυπνοι τρόποι. Να λυθούν τα προβλήματα, να δούμε γιατί τα προβλήματα αυτά προξύνονται. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ε, ακούσαμε από πλευρά κάτω χωρών. Εάν συνεχίσουμε τις ίδιε πολιτικές, τότε η κάθε χώρα σε πέντε χρόνια θα εξαρτάται ακόμη περισσότερο από τις προσδοκίες. επομένω. Α συνεργαστούμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μην έχουμε τέτοιου εξαρτήσεις στο μέλλον. Και να πιάνει πιο αποτελεσματική κοινωνική προστασία, κοινωνική πρόνοια σε όλες τις χώρες. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τα κρατημέλη. Απλώς η Ευρώπη σαν Ευρώπη όλοι μαζί θα προχωρήσουν προς τα εκεί. Ας κινηθούμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά την παρεμποδίουσα μειοψηφία. Ναι. Είναι δύσκολο και να ξέρει ακριβώ και όλα όσα γίνεται στι διαπραγματεύσει. Βέβαια, ξέρουμε ότι και η Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία παρεμποδίζουν. Οπότε είναι σοβαρό το θέμα. Εάν μία από τι δύο χώρε σταματήσει να παρεμποδίσει, αν δώσει το, το πράσινο φω, και ξέρω ότι λέγαμε στη Γερμανία, το κάναμε αυτό, το θεωρούμε ε, λάθος, ε, το βάλουμε πίσω μας και αυτά, ναι. Και, και εμείς θα θέλαμε να μην υπάρχει τέτοια κατάσταση, τέτοια ζήτηση, τέτοια ανάγκη. Αλλά τώρα έχουμε τριπλάσιους μειονεκτούντες, τριπλάσιους που έχουν ανάγκη από μια τέτοια πολιτική. Άρα είμαστε ρεαλιστές Το τελευταίο όσον αφορά τα διοικητικά να δούμε πώς μπορούμε με αυτό το πρόγραμμα να μάθουμε περισσότερα και επίσης το θέμα των πόρν θέλουμε το Κοινοβούλιο να βοηθήσει όλες οι οργανώσεις που ασχολούνται με αυτά τα προβλήματα ε, ε, ε, η πληγοδότησή μας συνέχεια συρρυκνώνεται δεν γίνεται να επιβιώσουμε στο μέλλον με την αρχή της φθήνουσας πρόοδου, της μειώσεως των πόρων. Ναι, όντως έτσι θα είμαστε ανεξάρτητοι, αλλά δεν θα υπάρχουμε. Υπάρχουν, υπάρχουν κάποιοι πυρογνώμονες που ξέρουν πώς μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους πόρους. Υπάρχουν λύσεις. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Μπέρτ. Δύσκολο σε πέντε λεπτά να απαντήσει, να απαντήσει κανείς όλες τις ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την, ε, το συσχετισμό με το κοινωνικό ταμείο. Καταλάβαμε ότι ξεφεύγουμε από την κοινή αγροτική πολιτική πλέον στην Ένωσή μας. Εάν και θεωρούμε ότι με τα πλεονάσματα της αγροτικής πολιτικής που μειώνονται αλλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν πιστεύουμε, εδώ Νομίζω ότι θα ήταν ε, χρηστή διαχείριση να ε, κατευθύνονται τα πλεονάσματα αυτά στο Ταμείο Ενίσχυσης των Πλέον Μενεκτούντων. Πάντως, καταλάβετε μας, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανταγωνισμό μεταξύ ενώσεων ή οργανισμών. Είμαστε ε, ανθρωπιστές που εργάζονται για ανθρωπιστικά δικαιώματα. Ε, δεν θέλουμε να κάτσουμε να κάνουμε ανταγωνισμό ποιανού το πρόγραμμα είναι το καλύτερο ή να λέμε ότι η δική μου, ο δικός μου σκοπός είναι ιερότερος από του διπλανού. Όχι, θέλουμε να επικεντρωθούμε στην επιχειριστική βοήθεια, ακόμα και αν υπάρχουν κάποια βασικά προϊόντα τα οποία πρέπει να ενισχυθούν, όπως αυτά για τους αστέγους και ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Σπίνεγουαν. Αλλά σε σχέση με τα ποσά, είναι σαφές ότι το ταμείο αυτό θα προσφέρει βοήθεια σε 27 κράτη πλέον από ό,τι 20 στο παρελθόν. Δύο ή 2,1 δις θα είναι η πρικοδότηση, ενώ θα έπρεπε να είναι 3,5 δις, δηλαδή είναι περίπου το μισό για χώρες που βρέθηκαν σε μια νέα κατηγορία και στο παρελθόν αποφελούνταν περισσότερο. Αυτό για τη Γαλλία αλλά και άλλες χώρες που θα μειωθούν περίπου στο ίμιση οι πόροι που τους διατίθεται. Αλλά εδώ και πέντε χρόνια ε, υπάρχει διαρκής μείωση. 50 εκατομμύρια ήταν η αρχική πρικοδότηση. Τώρα για τη δική μας την οργάνωση είχαμε 35% αύξηση των ανθρώπων που υποδεχόμαστε. Εάν πούμε ότι το 35% της αύξησης της δικής μας ε, χρηματοδοτήθηκε με μικρότερο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μείωση. Και εδώ μπορούμε να προσπαθήσουμε περαιτέρω με την πολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων, με την ενίσχυση των δημοσίων αρχών, με τη συμμετοχή των ελεγκτικών αρχών και να καταλάβουμε ότι έχει μειωθεί το ποσοστό της ευρωπαϊκής βοήθειας που διατίθεται στον καθένα ξεχωριστά. Εάν τώρα σταματήσει το 2014 το πρόγραμμα θα έχουμε 130 εκατομμύρια γεύματα λιγότερα στη Γαλλία. Δεν θα υπάρχει αντιστάθμιση αν σταματήσει αυτό. Δηλαδή 100 εκατομμύρια επαφές λιγότερες το χρόνο θα δημιουργηθούν, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες άτομα θα βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας δεν έχουμε εδώ κανένα μαγικό ραβδάκι, ούτε μπορούμε να προτείνουμε κάποια μαγική συνταγή. Αλλά ακόμα και με τη μείωση στο μισό, ακόμα και αυτό είναι μία ε, αλλαγή που δύσκολα θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε. Τώρα για τη λειτουργία και την ε, διαχείριση του προγράμματος. Εάν υπάρχει συγχρηματοδότηση από τα κράτη, θα πρέπει να σκεφτούμε πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, μπορούν κάποια κράτη με ιδιαίτερες δυσκολίες να μην ε, αναγκαστούν να περάσουν σε χρηματοδότηση για να μην μειωθεί και η βοήθεια, για τα πλέον ευάλωτα κράτη δηλαδή. Ε, ο κανονισμό βέβαια τα προβλέπει αυτά. Και για να μην είναι η ρύθμιση ιδιαίτερα περίπλοκη. Εμεί δεν είμαστε managers ακόμη και αν διαχειριζόμαστε πόρους οικονομικούς που μας έχουν διατεθεί εμείς, είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε, είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε σε ανθρωπιστικές οργανώσεις για να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους, όχι για να διαχειριζόμαστε χαρτοφυλάκια και κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν ότι θα πρέπει η αδειοδότηση, η, η προχρηματοδότηση να μην γίνουν δική μας αρμοδιότητα. Το πρόγραμμα το, στην προηγούμενη εκδοχή του υπάρχει εδώ και μία πενταετία. Δεν υπήρξαν ούτε ατασταλίες ούτε παρεκτροπές στη χρήση του προγράμματος. Υπήρχε ex post έλεγχος ο οποίος ε, ήταν επιτυχημένος. Δεν χρειάστηκε ποτέ να υποβάλουμε μία αίτηση, ένα φάκελο αίτησης πριν λάβουμε τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν οι απαντήση μου εντός πενταλέπτου. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κοστέλο, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φορείς ε, που ήρθαν ε, σήμερα εδώ. Αυτά που μας είπαν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα. Και επίσης ε, θέλω για, μια φορά, για άλλη μια φορά να στηρίξω αυτά που είπε ο κ. Σέκων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε στις επιτόπου, σε επιτόπια βάση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τα μέλη. Νομίζω η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Υπάρχουν αρκετές απόψεις που εκφράστηκαν και νομίζω θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε ε, ανακεφαλαίωση σε κάποια θέματα. Από τους φορείς αναφέρθηκε από την αρχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι πρόκειται για ένα ταμείο με μικρά ποσά δεν είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εξαλείψει τη φτώχεια. Παρόλα αυτά όμως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό να εκφράζει κοινωνική αλληλεγγύη με ανθρώπους που υποφέρουν από εξαθλίωση. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ε, αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Δεν λέμε δηλαδή ότι θα την εξαλείψουμε ή ότι θα επιληθεί πλήρως το πρόβλημα της φτώχειας. Νομίζω ότι αυτό ε, πρέπει να λεχθεί. Επίσης, ε, θέλω να συστήσω στους φορείς και σε όλους όσους συνάντησα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, συνάντησα μερικούς από αυτού και άλλε ιρλανδικέ οργανώσει και γνωρίζω πολύ καλά ότι το Ταμείο με την τρέχουσα μορφή του ίσω να είναι σταγόνα εν το ωκεανό, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, μπορείτε να δεχτείτε δωρέ, ε, ε, βοήθεια εθελοντών, ε, άλλα υλικά αγαθά, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ας έρθουμε τώρα σε κάποια από τα θέματα που τέτοισαν, όπως ε, παραδείγματος χάρη παραβιάζεται η αλληλεγγύη και η νομική της βάση. Νομίζω ότι υπάρχει μια νομική βάση για αυτό το πρόβλημα και αυτό ε, συμβαδίζει με αυτά που προβλέπει η συνθήκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευημερία όλων των πολιτών και συμβαδίζουν επίσης και με το στόχο που είναι η στρατηγική του 2020. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχει μια νομική βάση. Λαμβάνω βέβαια υπόψη μου τις ε, ε, επιφυλάξεις των εκπροσώπων σχετικά με τη χρηματοδότηση και δυστυχώς τα δυσάριστα νέα είναι ότι αυτή η Επιτροπή δεν μπορεί στις συστάσεις της να ζητήσει αύξηση κονδυλίων στον προεπλογισμό. Πάντως θα λάβουμε υπόψη μας αυτά που μας είπατε και θα προσπαθήσουμε όπου μπορούμε να σκίσουμε πολιτική επιρροή έτσι ώστε το ε, Ταμείο να έχει τα ελάχιστα απαραίτητα κονδύλια. Επίσης ε, θέλω να αναφερθώ λιγάκι στη συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι ένας ε, τομέας που μπορούμε να τον εξτάσουμε να μιλήσουμε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο, γιατί σας λέω, ήδη ε, γνωρίζουμε ότι ε, μοχλεύεται έτσι κι αλλιώς ε, τόσα πολλά κονδύλια. Αυτό που έχει σημασία... μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, ρωτάει ο μιλήτρια, ρωτάει. μιλάω γρήγορα γιατί νόμιζα ότι έχω μόνο πέντε λεπτά. Όσον αφορά το EFSF, νομίζω είναι σημαντικό ε, το ότι αυτό είναι ένα ξεχωριστό εργαλείο και ε, πρέπει λοιπόν ε, να επεκτείνουμε τους στόχους του. Θα μιλήσω στους σκιώδησηγητές για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα τους μιλήσουμε για το επίπεδο της ε, διαχείρισης έτσι ώστε η γραφειοκρατία να παραμείνει στο ελάχιστο. Η μεταφορά της γνώσης είναι πολύ σημαντική και αυτό είναι ένα από τα ε, συνοδευτικά μέτρα. Υπήρξε λοιπόν έκκληση να μην υπάρξουν πολλές αλλαγές στο πρόγραμμα γιατί είναι καλό. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν τομείς που μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Ε, τελείωσε, φτάνει, φτάνει λέει Πρόεδρος, ε, μετά, μετά. Ε, Δεν θα τα συζητήσουμε τώρα αυτά. Ε, είναι κρόαση αυτή. Να θυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Εξέτασε το σχεδίο έκθεση στις 21 Ιανουαρίου. 21 και 22 θα ψηφίσουμε. Η υποβολή τροπολογιών θα είναι πολύ σύντομη, διότι θέλουμε να παρακολουθήσουμε και τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό έξι ημέρες για την υποβολή τροπολογιών στις 26 ε, Φεβρουαρίου το μεσημέρι. 20 και 21 Μαρτίου θα εξεταστούν συμβαστικές προτάσεις στις 22 Απριλίου και την επόμενη μέρα θα ψηφίσουμε στο το Μάιο να περάσει από την Ολομέλεια η έκταση. Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει έτσι η συζήτηση με το Συμβούλιο. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε στο Μάιο να έχουμε φτάσει στην Ολομέλεια, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να ευχαριστήσω θερμά του πέντε προσκεκλημένους μας. Ναι, Ζητώντα συγγνώμη βέβαια για τον αυστηρό χαρακτήρα μιας ακρόασης, όπως συχνά συμβαίνει, αλλά ήταν σημαντικό στοιχείο να ακούσουμε τις συνεσφορές σας και να εμπλουτιστεί η έκθεση της εισηγήτριάς μας, η οποία νομίζω ότι μπόρεσε να αντλήσει την ουσία των παρεμβάσεών σας όταν εξεταστεί η έκθεση στις 20 Φεβρουαρίου είμαι σίγουρη ότι θα φροντίσει να απηχηθούν όλες σας οι παρατηρήσεις. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό στην σε διάταξη και περνάμε στο σημείο 16. Παρουσίαση του προγράμματος τεσσάρων εκθέσεων για τους οργανισμούς που αφορούν και το έργο της δικής μας Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη από τους διευθυντές μας, αλλά θα παραχωρήσω την Προεδρία στην Αντιπρόεδρό μας την κυρία Χίρς. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει από την κυρία Κρίστα Ζέλατσεκ, που είναι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Έχετε το λόγο για να μας κάνετε την παρουσίασή σας σε 7 λεπτά. Thank you very much uh, and thank you for the... Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δώσατε αυτή την ευκαιρία Να σα πω σε αυτέ τι να δώσω τη, τη γενική έποψη των τριών βασικών στρατηγικών θεμάτων που μα απασχολούν ε, ή μα απασχόλησαν μάλλον το 2012-2013, αλλά και για το μέλλον. Συγγνώμη, με την πρώτη διαφάνεια. Πρόκειται για αυτήν την, την, την, την καμπάνια για την υγεία στο, στην εργασία. Αυτό το κάναμε, το ξεκίνησε το 2012 ε, και συνεχίζεται ακόμα για να υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση του, του, της υγείας στην εργασία και οπότε και αυτή η εξτροετία αφορά επίσης τη συμμετοχή στη δουλειά, την, την, ιδιότητα του ε, και επίσης δέχομαι να ενθαρρύνουμε τους top managers να είναι πιο δραστήριοι όσον αφορά το, το, το, την προαγωγή αυτού του είδους των ε, των αρχών που θα μειώσουν τους κινδύνους της χώρου Μέχρι σήμερα αυτή μας ε, η εκστρατεία ήταν πάρα πολύ ε, ε, επιτυχής, γενικής φύσεως, αλλά πάντως καταφέραμε να έχουμε τα το τέλο υλικό. Σας ευχαριστώ. not functioning. No, I did. I did, yeah. You have to push forward. I push forward. maybe to use the seven minutes. Uh, Ariel. Α, πάντα 7 λεπτά. Α, όχι, εντάξει, εντάξει. Και επίσης αναπτύξαμε υλικό σε 24 γλώσσες και έχουμε επίσης μια σειρά από δημοσιεύσεις, ε, δίσκους, ε, φυλάδια και όλα αυτά μάλλον έχουν εκτιμηθεί. Όλα αυτά έχουν ε, σχέση με τον ρόλο των μάνατζερ και λοιπά. από αυτό το οποίο κάναμε συνδυάσαμε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα με άλλους φορείς και, μοιράσαμε το υλικό αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη και ίδια έχω συμμετάσχει σε πολλά από τα σεμινάρια που γίνανε και αυτά και στα, στα περισσότερα κράτη-μέλη αναπτύχθηκε δραστηριότητα και επίσης είχαμε δύο γύρους ε, προσλήψεων. Ε, είχαμε 85 εταίρους μέχρι σήμερα όλους αυτούς τους επιστρατεύσαμε τέλος πάντων και επίσης έχουμε μια σειρά από οργανώσεις κοινωνικούς εταίρους, πολυεθνικές και πανευρωπαϊκές οργανώσεις. Όπως πάντα υπάρχει και αυτό το έπαθλο για την καλύτερη πρακτική και έχουμε 50 αιτήσει από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη και έχουμε μια διαδικασία επιλογής. Οπότε έχουμε 10 ουραδευθέντες και 10 επενεθέντες. Πάρα πολύ θετικά όλα αυτά. Συνάντηση κορυφή θα γίνει στο Μπιλμπά τον Νοέμβριο του 2013. Θα συνδιοργανωθεί με την Λιθουανική Προεδρία. Αρχίσαμε να οργανώνουμε την επόμενη εξοδία μας. Το θα Ασφάλεια και Υγεία Εργασία υπαριθμών 3. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στις εταιρείε και συμβολή από κοινωνικούς εταίρους και κράτη-μέλη. Από ό,τι φαίνεται, τα κράτη-μέλη εκτιμούν το έργο μας. Άλλο. Άλλο μέρος που θέλουμε να θέξουμε... είναι η ανάπτυξη ενεργής εκτίμησης του κινδύνου μέσω ίντερνετ για τις επιχειρήσεις. Το λέμε όριο αυτό το πρόγραμμα και αυτή η δραστηριότητα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Και όλο ένα και περισσότερα κράτη-μέλη τώρα συμμετέχουν. Έχουν το δικό τους πρόγραμμα όριο σε εθνικό επίπεδο, σε τομεϊκό επίπεδο και μετά την περίοδο της δοκιμής Προχώρησαν παραπέρα. Τον Ιούνιο του 2012 έγινε η γενική δοκιμή. Όμως τώρα θα υλοποιήσουμε την ε, περαιτέρω εξέλιξη του προγράμματος. Πολύ πρακτικό αυτό για την εκτίμηση του κινδύνου μέσω του ίντερνετ. Ήδη έχουμε πορεύσει νέα μνημόνια με τα κράτη-μέλη και ακομα περισσότερο περισσότερα κράτη-μέλη έχουν αρχίσει τις επαφές για να χρησιμοποιήσουν σε εθνικό επίπεδο αυτό το πρόγραμμα. Σαν χιόνο στη βάδα Όλο ένα και περισσότερα κράτη-μέλη μπαίνουν στο παιχνίδι. Συνεργαζόμαστε επίσης με εθνικού φορείς και τουλάχιστον 8 τομιακοί κοινωνικοί εταίρε συνεργάζονται και αναπτύσσουν το δικό του λογισμικό όριο. Και βέβαια η υπηρεσία μας βοηθά για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη, κατάρτιση, παροχή βοήθειας. Πρόκειται για ένα από τα βασικά θέματα, ότι θα τέτοιου είδους ε, εργαλεία να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν να απορροφήσουν τη χρηματοδότηση, να μοιράζουν παντού οδηγίες και τα κρατημέλη να μπορούν να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση που υπάρχει και έτσι αυτό το διαδραστικό μέσο να αξιοποιείται. Τώρα τελευταίο τομέα δραστηριοτήτων έχει σχέση με δεν τα καταφέρνω καλά. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό αφορά με κάποιο πρόγραμμα που ξεκινήσαμε σε σχέση με τους πιο ηλικιωμένους, ε, μεγαλύτερους εργαζομένους σε σχέση με την υγεία στο χώρο της υγείας και έχουμε τώρα αυτή τη δράση που χρησιμοποιεί, που αξιοποιεί ένα κονδύλιο 2 εκατομμυρίων. Έχουμε κάνει δύο εκθέσεις για το δίκτυο 15 προβλέπεται μια διάσκεψη και θα, θα διερευνήσουμε, θα δούμε αυτό, αυτό το πρόβλημα που λέγεται όσπας, πώς τα πάει, τι έχει γίνει σε επίπεδο κράτου μέλους, σε επίπεδο λογιάς. Θα διαδώσουμε μόνο στα σχετικά εργαλεία και θα δώσουμε δημοσιότητα σε κάποια συμπεράσματα θα συνεργαστούμε την ίδια για την Απασχόληση και επίση θα σας διαβάσουμε και κάποιες συστάσεις. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα αναφέραμε το πρωί. Να διευρυνθούν οι στρατηγικές και τα προγράμματα μπορούν να, να, να, να βελτιώσουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων και κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία. Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική που την έχουν καλλιάσει τα κράτη-μέλη. Το Δεκέμβριο σημειώθηκε συμφωνία και ελπίζουμε ότι η σχετική στρατηγική που συμφωνήθηκε τότε ελπίζουμε το 2013 να αποκρισταλωθεί. Και βέβαια αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ελπίζουμε να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική ως και έτσι ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με την Επιτροπή. Αν έχετε ερωτήσει να τις απαντήσω. Αλλά ε, να δούμε και με αυτή τη συμφωνία που είπαμε το πρωί. Ναι, είναι σημαντική η συμφωνία που είναι για την έδρα μας στο Μπιλμπάο. Θα προσυπογράψει η Ισπανική Κυβέρνηση το σχετικό κείμενο έχει αποκρισταλωθεί, αλλά βέβαια επειδή πρόκειται για διεθνή συνθήκη, διεθνή συμφωνία, ε, παίρνει κάποιο χρόνο. Ευχαριστούμε κυρία Στέντλατσεκ και τώρα κύριο κύριος που είναι διευθυντής του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή επασχόληση για την υποστήριξη του κέντρου μας και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε το 2011. Όπως ξέρετε, το κέντρο μας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πρόσληψη νέου διευθυντή, ε, καθότι οι δύο προηγούμενες ε, διαδικασίες αποδείχθηκαν άγονες. Σε αυτή λοιπόν τη φάση θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω την κυρία Προύσα που έχει οριστεί από τον Νοέμβριο του 2012 ε, ως ε, διευθύντρια που ενεργεί χρέη διευθυντού. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, καθυστερεί περαιτέρω και κυρίως η ανέργηση του κτηρίου γιατί υπάρχει ε, γεωλογικό πρόβλημα το 2011 ε, καταρτίστηκαν προγράμματα μέχρι το 2013 και ένα λεπτομερές πρόγραμμα το οποίο ε, είναι ε, διαθέσιμο στην ισοσελίδα. Τώρα, το πρόγραμμα εργασίας του 2012 εφαρμόστηκε επιτυχώς. Ε, επίσης, ε, χρησιμοποιήσαμε ε, τις, τα κονδύλια που μας εντόθησαν, άρα δηλαδή πλέον δεν υπάρχουν άλλα αποθέματα. Και αποδείχτηκε και η ε, καλή λειτουργία του κέντρου μας. Το 2013 ο αγώνας ε, κατά της ανεργίας των νέων ε, και η απόκτηση καλύτερων δεξιοτήτων όπως επίσης και η μεταρρύθμιση των συστημάτων για να διασφαλίζεται η διαφάνεια, αυτά έμειναν στο επίκεντρο της ε, δικής μας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν τα εξής ποσοστά. 46% ε, ε, χωρίς πολλές ιδιότητες, ένα αρκετά μεγάλο ποστό, 50% με τρία κατάρτιση και το 10% ε, πανεπιστημιακή κατάρταση. Αυτό ήταν παλιά η αναλογία. Τώρα όμως 40% πανεπιστημιακή κατάρτιση και 10% είναι μόνο αυτή με τα πολύ περιορισμένα προσόντα. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Ε, σημαίνουν ότι η ε, μεσαία εκπαίδευση εξακολουθεί να επικρατεί, άρα δηλαδή εδώ υπάρχει ένα δυναμικό περαιτέρω ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Βέβαια έχει αλλάξει και η δομή ε, των ε, άμεσα ενδιαφερόμενων και δεν εκπλήσει το γεγονός ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία βέβαια ελήφθησαν από διάφορες χώρες για να ε, βελτιωθεί η κατάσταση για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και να μπορέσουν και εκείνοι να ολοκληρώσουν με μια μεσαία, με μεσαία προσόντα. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στην Αυστρία, ας πούμε, για να ε, μπει κανείς σε μαθητεία πρέπει να είναι 14 ετών. Τώρα στη Γερμανία είναι πάνω από τα 16 για να ξεκινήσει κανείς ε, μαθητεία. Και έτσι λοιπόν πάνω στο, ε, στον εξής συλλογισμό. Βλέπουμε ότι η κατάρτιση έχει μεγάλη σημασία για την ανεργία των νέων. Ελέγξαμε την κατάσταση και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες χώρες που αντέδρασαν σε αυτό το έγγραφο. Ε, αργότερα υπογράφηκε ένα μνημόνιο ανάμεσα στη Γερμανία και έξι άλλες χώρες όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να ελέγχονται οι δραστηριότητες. Και βεβαίως εκεί συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ε, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ε, μαθητεία για να λυθεί το πρόβλημα και ε, να εξευρεθεί τουλάχιστον κάποια λύση για τα πολύ ψηλά επίπεδα ανεργίας νέων που ε, βιώνουμε σε κάποιες ε, χώρες. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ε, στη Θεσσαλονίκη για το 60% των νέων. Υπάρχουν νέες προδιαγραφές και νέοι όροι για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ε, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, θα προσφέρει ε, στοιχεία για να γίνεται καλύτερος έλεγχος της διαδικασίας της Κοπενχάγης συστάσεις που να αφορούν συγκεκριμένα κάποιες χώρες. Πέρυσι εδώ πάλι ανέφερα ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε εξοικονομήσεις. Σας είπα με το παράδειγμα ότι περιορίζουμε τις αποστολές, κάνουμε πολλές video conference, χρησιμοποιούμε το Skype για να κάνουμε τις συνεντεύξεις στη διαδικασία των προσλήψεων. Ε, πάντως η κατάσταση είναι η εξής. Ήδη τώρα ε, το κέντρο ζητάει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου γιατί χρειαζόμαστε και άλλους πόρους για το 2014. Ε, αυτά συζητούνται αυτή τη στιγμή μεταξύ Επιτροπής ε, και Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και όμως μόλις έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο θα σας κατατεθεί με σίγουρος και θέλουμε να μπορούμε να υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ κύριε Λετμαγερ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μενέντες Φαλέντες τώρα, που είναι πρόεδρος του Eurofund. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ελπίζω να λειτουργεί ο προβολέας. Το μηχάνημα των slides. Ήθελα να μιλήσω για το Eurofund και το 2012 ολοκληρώθηκε το τετρατές μας πρόγραμμα. Διαβίωση και ευκαιρίες για όλους. Ξεκινάμε το... τη νέα φάση του προγράμματος για το 2013-2016. με πλέον τεκμηριωμένες πολιτικές για ισχυρότερη Ευρώπη. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο λοιπόν και δεν θα σα παρουσιάσω όλε τι λεπτομέρειε, αλλά κάποια από τα σημαντικότερα σημεία αυτού του τετραετούς προγράμματο. Κάποια από όσα δεν θα θίξω θα τα δείτε και στα έγγραφα που θα αφήσω στην αίθουσα φεύγοντα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε τομεί όπου έχουμε ιδιαίτερε τεχνικέ γνώσει και έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι συνθήκε εργασία, η βιομηχανοποίηση και ο κοινωνικό διάλογο, οι συνθήκε διαβίωση και οι διαρθρωτικές αλλαγές καθώς και αναδιάρθρωση. Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας θα βασίζεται στις εργασίες παρακολούθησης όπως γινόταν ως τώρα. Οι περισσότεροι γνωρίζετε τις τρεις υπηρεσίες που διαχειριζόμαστε. Την μελέτη για τις ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίες, για την ποιότητα στην αγορά εργασίας και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Σε 34 χώρες εκπονούνται οι μελέτες αυτές και η συνοπτική έκθεση λόγω χάρη για τις συνθήκε εργασία, αν θυμάστε, παρουσιάστηκε το 2012 σε αυτό το κοινοβούλιο, μάλιστα, με παρουσία του Προέδρου Μάρτιν Σούλτ, σε μια διάσκεψη όπου συζητήθηκε το θέμα της ποιότητας ε, στην εργασία. Η μελέτη για την ποιότητα στην εργασία παρουσιάστηκε στο τέλος του 2012 επίσης, με τα βασικά της πορίσματα εδώ στις Βρυξέλλες, ενώ για τις ευρωπαϊκές εταιρείες θα έχουμε παρουσίαση στις αρχές της φετινής χρονιάς. Μπορείτε στον ιστότοπό μας να δείτε χαρτογράφηση των μελετών που ως τώρα έχουν εκπονηθεί. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση αναχώρα ε, και να βρει συγκεκριμένα στοιχεία. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέρος των δραστηριοτήτων παρακολούθησής μας ε, οφείλονται και έχουν ε, συγκεντρωθεί χάρη στα παρατηρητήρια που έχουμε, παρατηρητήριο για τις συνθήκες εργασίας και άλλα δύο. Με το νέο τετραετές ε, πρόγραμμα θα ενσωματωθούν σε ένα τα τρία αυτά παρατηρητήρια για τις συνθήκες του επαγγελματικού βίου. Επίσης έχουμε και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Αλλαγών. Μετά την Σύνοδο της Νίκης δημιουργήθηκε, αν θυμάστε, το 2001. Συνδυάζουμε τα πορίσματα των ερευνών μας με πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω των Ευρωπαϊκών Παρατηρητηρίων και ενδελεχείς μελέτες. Τα τελευταία χρόνια επικεντρωθήκαμε σε πτυχέ που είχαν να κάνουν με τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης ιδιαίτερω. Να τονίσω τρία παραδείγματα από τα πορίσματά μας σε σχέση με τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης. Πρώτον, τα πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα του τρίτου, της τρίτης μελέτης για την ποιότητα της ζωής που κάναμε σύγκριση των στοιχείων πριν και μετά την ε, έρευνα. Ένα τρίτο των Ευρωπαίων πολιτών ανέφεραν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Βλέπετε ότι είναι μεγάλη η δυσκολία να τα βγάλουν πέρα οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά αυτό ξεκινάει από ένα 22% στην Ελλάδα με ένα πολύ μικρό ποσοστό στη Φινλανδία μεγάλη ποικιλομορφία. Το επίπεδο αισιοδοξία, ικανοποίηση από τη ζωή των ατόμων έχει μειωθεί 20% σε κάποια κράτη-μέλη. Βεβαίω τα κράτη-μέλη αυτά είναι αυτά που έχουν πληγεί κατεξοχήν από την κρίση. Η Ευρώπη είναι ένα καλό τόπο διαβίωση, μεν, αλλά η κατάσταση δυστυχώ έχει επιδεινωθεί. Βεβαίω αυτό που πλέον ανησυχεί του πολιτικού ευθύνοντες και εσά φαντάζομαι του βουλευτέ είναι η πτώση του ποσοστού εμπιστοσύνη προ τα θεσμικά όργανα, ιδίω τι κυβερνήσει και τα κοινοβούλια. 4,1 για τα κοινοβούλια και 4 για τι κυβερνήσει σε μια κλίμακα του 10. Όμω υπάρχει και μεγάλη απόκληση στα αποτελέσματα μεταξύ των κρατών μελών. Αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό βαθμό. Η κρίση έχει πλήξει κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, περισσότερο από ό,τι άλλες δηλαδή, τους νέους ας πούμε, όπου βλέπουμε τι γίνεται με τους νέους το δεύτερο παράδειγμα. Θα θυμάστε με την έκθεση που δεσμεύσαμε φέτος, καθώς επικεντρωνόμασταν περισσότερο στους νέους, κοιτάξαμε τι γίνεται με αυτούς που αποκλείονται από την εκπαίδευση, ε, την κατάρτιση και την τεχνική εκπαίδευση, τους λεγόμενους NITS, ε, ένα τρί, 14 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 14,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού μεταξύ 15 και 29. 1,2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ χάνεται εξαιτία αυτού του φαινομένου. 153 δι το 2011. Ακόμη πιο σημαντικό το γεγονό ότι Υπάρχει και κοινωνικό κόστος, για το οποίο πραγματοποιούμε μελέτη και θα την παρουσιάσουμε σύντομα. Απαιτούνται μάλιστα συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα για να αναχαιτευτεί αυτό το φαινόμενο. Τρίτο παράδειγμα, ο αντίκτυπο της κρίσης. Συνέπειες της αναδιάρθρωσης. Μελετήσαμε τις πιθανότητες και το προφίλ των ανθρώπων που μπορεί να χάσουν τη δουλειά του. Συγκεντρώσαμε δηλαδή τα χαρακτηριστικά αυτών που έχουν σοβαρέ πιθανότητε να χάσουν τη δουλειά του. Και μάλιστα έχουν λίγε πιθανότητε να βρουν άλλη θέση. Αλλά επικεντρωθήκαμε και σε όσου παραμένουν σε αναδιορθωμένε εταιρείε οι επιχειρήσει. Αυτέ οι εταιρείε προσπαθούν να γίνουν ανταγωνιστικότερε, αλλά και οι εργαζόμενοι αυτοί απειλούνται από κοινωνικο-ψυχολογικού κινδύνου. Χρειάζεται και από αυτούς κάποια πολιτική, και για αυτούς κάποια πολιτική μέρημνα. Τώρα για το νέο τετραετές πρόγραμμα. Έχουμε το στόχο να παρέχουμε υψηλής ποιότητας επίκαιρα και πολιτικά εύστοχα δεδομένα για τους πολιτικούς ηθήνοντες, επικεντρωνόμενοι σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας. Πρώτον, ε, για τις αγορές εργασίας και την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με παραδείγματα όπως το, την παρακολούθηση της δουλειάς, της αλλαγές, ε, της τα χαρακτηριστικά της εργασίας, την ποιότητα της εργασίας ή το μέλλον, τη, το τομέα του βιοτεχνικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα οι συνθήκες εργασίας και τι συνθήκε απαιτούνται για να είναι βιωσιμότερη η εργασία, εφόσον θέλουμε να δουλεύουν περισσότεροι εργαζομένοι. Έπειτα οι βιομηχανικέ σχέσει σε μεταβαλλόμενα πολιτικά τοπία. Λόγου χάρη οικονομική διακυβέρνηση, μισθολογική κλίμακα και γενικότερε επιπτώσει και έπειτα τα πρότυπα διαβίωση, προδιαγραφέ διαβίωση και κοινωνική συνοχή. Κοινωνικέ υπηρεσίε όπω η φροντίδα των παιδιών, η υγειονομική περίθαλψη, ή το τι γίνεται με τους νέους και την ενσωμάτωσή τους. Αυτό που θέλουμε είναι να παράσχουμε πληροφορίε ώστε να υπάρχουν καλύτερα τεκμηριωμένε πολιτικέ αποφάσει. Ε, μελετώνται όμω και οι επιδόσεις μα για να δούμε κατά πόσο οι δικέ μα συνεισφορέ χρησιμεύουν στου πολιτικού ευθύνοντε. 204 πολιτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκαν στα πορίσματα της ε, Eurofund το 2012. Εδώ έχετε κάποια παραδείγματα, 29 ευρωπαϊκά έγγραφα του Κοινοβουλίου. Κάποιοι τα γνωρίζουν από την Επιτροπή σας, όπως η έκθεση για την πληροφόρηση και την διαβούλευση με εργαζομένους στην πρόληψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων ή η έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ή άλλε εκθέσει που έχουν συζητηθεί σε άλλε επιτροπέ, όπω την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών, για τι συνθήκε εργασία των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών ή τον αντίκτυπο τη οικονομική κρίση στη δημιουργία, το δυναμικό ε, δημιουργία θέσεων εργασία στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Επίση και σε έγγραφα τη Επιτροπή, όπω η εμβληματική έκθεση τη Γενική Διεύθυνση ε, ε, Επιχειρήσει για την οικονομική και κοινωνικέ εξελίξει στην Ευρώπη το 2012. σε αυτή την έκθεση και σε άλλους μας αναφέρουν διαρκώς και παραπέμπουν στα περιορίσματά μας όπως και σε έγγραφα του Συμβουλίου. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα τα οποία δεν προλαβαίνω να σας παρεθμίσω τώρα. Κάποια αριθμοί τώρα για να έχετε και κάποια εικόνα για το τι κάλαμε το 2012. Χρήση του προπολογισμού κατά 99% με το πλεόνασμα που προβλεπόταν για τις υπηρεσίες παρά την εκκρεμωδικία του ΔΕΚ με 97% λοιπόν ποσοστό θα είχαμε ξεκινήσει. Ο προπολογισμό μα ήταν 20.544.000, 172 δημοσιεύσει σε 831 γλωσσικές εκδοχές 100.000 downloads έγιναν περίπου από τον ιστοτοπό μας και 2 εκατομμύρια σχεδόν χρήστες επισκέφτηκαν τον ιστοτοπό μας. Εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις, με μεγάλη χαρά να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο, στη Μαντλίν Σάμπαλ της, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτης και παρακαλώ πολύ να παραμείνετε στα 7 λεπτά. Αυτή είναι η μοίρα πάντα του τελευταίου μιλητή. ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης για ε, την ε, πολύ σημαντική υποστήριξη που μας προσφέρατε κατά τη διάρκεια του 2012. Μια δύσκολη χρονιά και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό θα σας παρουσιάσω τις ε, βασικές μας ε, δραστηριότητες. Το 2012 ήταν, μια, ήταν η χρονιά εκείνη όπου στις χώρες της ε, Νότιας Μεσογείου η κατάσταση εξακολούθησε να είναι πολύ μεταβλητή. Εμείς λειτουργούμε για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτό στις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στις υπόλοιπες. Γιατί δραστηριοποιούμεθα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι η Ευρώπη θεωρεί ότι μπορεί να είναι πιο ισχυρή μόνο αν είναι ισχυρή ε, και ε, αν είναι ισχυροί οι γείτονες. Ε, πραγματικά θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις στις διάφορες αυτές τις περιοχές. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε και εδώ μιλάω για την ε, υπηρεσία που είναι υπό του διευθυντή που βρίσκεται στην Άτσο. Έγινε λοιπόν μια αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό της αναφέρει ότι το δικό μας το Ίδρυμα αξιολογήθηκε ως ε, ένα Ίδρυμα που συνεισφέρει ε, σημαντικά, προσφέρει προστιθέμενη αξία στις ε, παρεμβάσεις του και επίσης στην αξιολόγηση αναφέρεται πόσο σημαντικές είναι οι δραστηριότητές μας ε, για τις ε, ανάγκες των χωρών που σας ανέφερα. Το 12 λοιπόν συνεχίσαμε τη διαδικασία του Τωρίνου και με μεγάλη μου χαρά αναφέρω ότι η διαδικασία της Κοπενχάγης για την οποία είναι αρμόδια το ΣΕΝΤΕΦΟΠ η διαδικασία αυτή ε, είναι έμπνευση για μας ε, για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις χώρες εταίρους. Η διαδικασία του Τωρίνου για δεύτερη φορά εφαρμόζεται. Εξαίρεση λοιπόν από τη συμμετοχή, εξαιρέσει είναι πάρα πολύ λίγες για καθαρά πολιτικούς λόγους και θα καταλάβετε βέβαια γιατί η Συρία δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε και η Αλγερία και η Ισλανδία γιατί είναι μία από τις χώρες εταίρους ε, που παραμένει σε συνεργασία με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Αυτό που πρόκειψε καινούργιο το 2012 στη διαδικασία του Τωρίνου είναι ότι το Μάιο θα ολοκληρώσουμε μια, ένα μεγάλο συνέδριο και εδώ μας προσφέρεται η δυνατότητα να έρθετε όλοι ε, στο Τωρίνο και να δείτε την πραγματικότητα που υπάρχει στις διάφορες χώρες. Αυτά θα τα παρουσιάσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Το 2012 λοιπόν προσθέσαμε την διάσταση της governance, της η ε, απασχόληση δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο ένα ε, θεσμό. Είναι ένας τομέας πολιτικής που είναι το σταυροδρόμι διαφόρων τομέων και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτική, κοινό όραμα, κοινή εφαρμογή. Αυτό είναι το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή των διαφόρων στόχων της πολιτικής. Και αυτό είναι ο λόγος γιατί επίσης εισαγάγαμε τη μεθοδολογική υποστήριξη για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διότι εμείς, ε, όπως ε, σας είπα, ε, έχουμε σε οριζόντιο επίπεδο όλοι τα ίδια οράματα και επίσης διότι θεωρούμε ότι το πολυεπίπεδο πρέπει να ισχύει και για τις κοινότητες και για τις κεντρικές κυβερνήσεις. Ε, οι περισσότερες χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι συγκεντρωτικές και χρειάζονται τη βοήθεια σε τοπικό επίπεδο για να μπορούν να εκφράζουν τις διάφορες παρεμβάσεις τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ένας άλλος τομέας όπου δραστηριοποιηθήκαμε ιδιαίτερα το 2012 όπως συστήνει η διαδικασία του Τωρίνου είναι η επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι επίσης καθοριστικό σημασίας ε, για τις χώρες αυτές. Η ε, ανεργία των νέων ή των γυναικών είναι πάρα πολύ ψηλέ στις χώρες αυτές. Παράδειγμα, η Αίγυπτος που ε, παρουσιάζεται και στη δουλειά μας. Στην Αίγυπτο η δημογραφική έκρηξη θα λάβει χώρα ταχύτατα. Τα επόμενα 15 χρόνια θα χρειάζονται 35 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει έστω και μία χώρα στον κόσμο που να μπορεί να προσφέρει όλες αυτές τις θέσεις εργασίας. Όμως οι χώρες μπορούν να προσφέρουν ε, τα απαραίτητα προσόντα στους νέους έτσι ώστε μόνοι τους να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους. Ε, ποια είναι τα καλά νέα μετά από δική μας παρέμβαση, τουλάχιστον την περασμένη εβδομάδα στην Αίγυπτο η απόφαση ε, αποφάσισε να συστήσει ένα κεντρικό συμβούλιο. Δηλαδή, αντί οι επιχειρήσεις ε, να υπάγονται σε 23 υπουργεία, πλέον να υπάρχει συντονισμός, τουλάχιστον όσον αφορά την απόκτηση προσόντων σε μια χώρα με μεγάλη ανεργία. Και ένα άλλο στοιχείο λένε ότι η εδαφική έλλειψη συνοχής είναι πολύ μεγάλη γιατί ε, στο 8% του εδάφους, της, εδάφους τους είναι συγκεντρωμένοι οι Αιγύπτιοι. Άρα δηλαδή η συνοχή είναι επίσης ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες όπου οι συνάδελφοί μας ε, θα πάνε στην Αίγυπτο να συζητήσουν για τη διαδικασία του Τωρίνου γιατί το 2013 εκεί θα εφαρμόσουμε την διαδικασία του Τωρίνου λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Μία άλλη χώρα όπου κατ' το 2013 θα εφαρμόσουμε διαδικασία Τωρίνου είναι η Λιβύη, η οποία προσθέθηκε σε εμά το 2012 ε, δηλαδή τότε που είχα έρθει εδώ και σας παρουσίασα τις ε, δραστηριότητές μας. Είμαστε λοιπόν ο μοναδικός ε, ευρωπαϊκός φορέας, γραφείο, πέστε το όπως θέλετε, που δραστηριοποιήθηκε στη Λιβύη το 2012. Πολύ καλό αυτό, διότι το ανθρώπινο κεφάλαιο ήταν η μητέρα των προτεραιοτήτων όταν αρχίσαμε να ασχολούμεθα με την ανοικοδόμηση της Λιβύης. Όχι ότι σταμάτησε η διένεξη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τη χώρα αυτή η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι καθοριστική. Επίσης, το 2012 είχαμε και άλλη μια ευκαιρία ως οργάνωση να οργανώσουμε τον πολιτικό διάλογο ε, σε περιφερειακό επίπεδο. Και εδώ επιθυμώ να εκφράσω ε, θερμά την Επιτροπή Απασχόλησης και κυρίως ε, την πρόεδρό της, έστω και αν λείπει, ε, διότι υποστήριξε την ε, συνάντηση των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας στο ΑΜΑΝ. Στο ΑΜΑΝ λοιπόν ελήφθη η απόφαση ότι ε, από τώρα όχι μόνο οι κυβερνήσεις θα προσκαλούνται για να συζητάνε πολιτικές αλλά και άλλοι παράμετροι. Και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε την υποστήριξή σας για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τα κοινοβούλια αυτών των χωρών έχοντας κατά νου ότι στα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχει ούτε ένας φορέας ή μια επιτροπή που να ασχολούνται με την απασχόληση και την κατάρτιση. Άρα δηλαδή χρειάζονται τη βοήθειά σας και εκείνοι και εμείς για να μπορούμε να συζητάμε για χάραξη πολιτικής, αυτό να το συζητάμε με θεσμούς που δεν έχουν ακόμα τις γνώσεις να αξιολογούν τι ακριβώς χρειάζεται η χώρα και το 2012 και δεν θα αναφέρω άλλα παραδείγματα ήταν επιτυχημένο ε, και από διοικητική σκοπιά και η έκθεση, ετήσια έκθεση πεπραγμένων που θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο ε, θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες. Εγώ θέλω απλά να πω ότι το 2012 με ένα προϋπολογισμό που ήταν κατά 1% χαμηλότερος από το 2011 κατορθώσαμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας και όπως σας είπα και να περάσουμε και σε μια νέα χώρα στη Λιβύη. Ελπίζω όμως ότι την επόμενη χρονιά θα γίνει η καλύτερη αξιολόγηση της κατανομής των πόρων και το 2014 δεν θα είναι η χρονιά εκείνη όπου ε, θα τεθεί ένα αμφιβόλο η ε, αξία του φορέα του δικού μας. Το 2014 θα είναι η χρονιά όπου θα προχωρήσουμε ε, και Έχω τη χαρά να αναφερθώ στους Πάρκιν και Άντερσον γιατί μιλάω για το πρόγραμμα εργασίας του 2013 που ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Νοέμβρη. Το 2013 θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα ε, για τα προσόντα σε συνεργασία με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Θα συνεχίσουμε την επαγγελματική κατάρτιση στην Ανατολική Ευρώπη. Εκεί οι ανάγκες των χωρών είναι παρεμφερείς και θα συνεχίσουμε και τη δουλειά μας όσον αφορά την απόκτηση προσόντων στη Μεσόγειο και άλλα δύο προγράμματα που θα σας τα αναφέρω. Η υποστήριξη στη Μεσόγειο ε, σε σχέση με την αντιμετώπιση της απασχολησιμότητας, κυρίως των νέων και των γυναικών. Και ένα άλλο πρόγραμμα που θα στηρίζει πιο ουσιαστική βοήθεια που θα δείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες της διεύρυνσης. Ε, Έχουμε λοιπόν τα οράματα του 2020 και αυτή θα είναι η στρατηγική η οποία θα συμφιλειώσει τις προτεραιότητες ε, σε πολλές χώρες. Ελπίζουμε, όπως σας είπα, η βοήθειά μας θα είναι πιο αποτελεσματική, πιο ουσιαστική. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της οικονομικής και κοινωνικής ε, ανάπτυξης ε, σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Όπω γνωρίζετε, λέει ο πρόεδρο, έχουμε τρει εμπειρογνώμονε, του οποίου έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίση και ε, το, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο τη Εκπαίδευση. Βρίσκονται εδώ και άρα του δώσουμε το λόγο. Ο καθένα για τρία λεπτά. Okay, I'm happy. I will speaking my... Ναι, εντάξει. Εντάξει, μου αρκεί και θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, ακριβώς όπως ε, όταν ήμουν εδώ. Να σας τα πω στα σουηδικά. Επέστρεψα λοιπόν και... Και ξέρετε, με επέλεξαν ως εμπειρογνώμονα. Λέω ο κύριος Άντερσον, διότι ήξερα πολλά για το ETF, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελμής εκπαίδευση. Και οφείλω να σας πω ότι όταν κανείς γίνει manager, μαθαίνει περισσότερο από όσα ήξερε πριν, γιατί ξέρει τις λεπτομέρειες. Δεν είναι θέμα το, το, το, τι λέγεται στα διοικητικά συμβούλια. Το πιο σημαντικό είναι η προετοιμασία. Εμείς λοιπόν οι εμπειρογνώμονες που μας καλέσατε και μας ορίσατε να μιλήσουμε σήμερα εδώ, έχουμε ασχοληθεί δραστήρια με τα προγράμματα, με την προετοιμασία των συνδυάσεων του Διευθυντικού Συμβουλίου και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ε, πολύ πολύ σημαντικό είναι τη δουλειά μας. Κοιτάξτε να σας πω δύο-τρία λόγια. Ε, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ το έργο το οποίο τώρα επιτελείται. Δεν ήξερα ότι γίνονται τόσο πολλά εκεί στο Ίδρυμα και ε, να σας πω τι άλλο με έχει ε, εντυπωσιάσει ότι ο κόσμος τα καταφέρνει να κάνει αυτά τα οποία του, ο καθένας κάνει αυτά που του έχουν ανατεθεί παρά το ότι υπάρχει συρρήγνωση του προπολογισμού παρά το ότι έχει συρρήγνωθεί το προσωπικό όμως παρόλα αυτά δεν έχει συρρήγνωθεί δεν έχει μειωθεί η δουλειά που πρέπει να κάνουμε μιλούμε για τις χώρες που Α αναθέτουν όλο ένα και περισσότερη δουλειά, γιατί προσπαθούν και αυτοί στο εθνικό επίπεδο να βελτιώσουν τι επιδόσεις του στον τομέα μας. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι η ευελιξία. Ακούσατε τι έγινε στην Αίγυπτο, στην ε, Λιβύη. Το γεγονός ότι το Ίδρυμα κατάφερε να συνεχίζεται ο διάλογος. Κατάφερε να επιστρατεύσει κάποιους πόρους και να στήσει κάποια πράγματα σε Αίγυπτο και Λιβύη. Ε, δηλαδή, το σύστημα προτιμούμε προσπαθούμε να, να λειτουργεί πάντα στις δυσκολίες που υπάρχουν. Προσπαθούμε ε, να προωθήσουμε μια καλύτερη συνεργασία παντού στην Ευρώπη. Μέσα στην παιδεία. Μέσα στην Ευρώπη. Με τις γειτονιάζουσες χώρες. Αυτό είναι ένα όραμα μακρόπνο. Δεν γίνεται ε, από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλουμε να έχουμε επαφές, θέλουμε να έχουμε κάποια συστήματα τα οποία να μπορούν να λειτουργήσουν μακρόπνοα. Και εσά ξέρουμε η προσέγγιση τέτοια είναι. Ελπίζουμε επομένω αυτό θα συνεχίσει στο μέλλον. Και έτσι λοιπόν προσπαθούμε να κινηθούμε, να μην έχουμε αλλαγές κάθε χρόνο, να συνεχίσουμε μια τέτοια προσέγγιση μακροπρόθεσμη, μακρόπνοη. Έτσι να δουλεύουμε. και σας ευχαριστώ που με καλέσατε και τώρα ε, να δώσουμε τη σκητάλη στη Σάρα, που δίπλα μου, η οποία είναι πιο παλιά από μένα στη δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη τριετή θητεία μου εδώ ως ε, εμπειρογνώμων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος αυτού. Δεν έχουμε ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ε, έχουμε δεσμευτεί και είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι ε, για λογαριασμό σας εκεί δίνουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας ε, να μην επαναλάβω όσα προελέχθησαν αλλά να δούμε τι γίνεται με αυτή την εξωτερική αξιολόγηση η οποία ήδη αναφέρθηκε πάρα πολύ καλά είναι όσα αναφέρθηκαν εκεί και είπαμε όμως ότι εδώ και τέσσερα χρόνια ασχολούμαι και βλέπω τις αλλαγές, βλέπω τις βελτιώσεις αυτή την περίοδο και Βεβαίω ε, δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε ε, περήφανοι και να έχουμε αυτοπεποίθηση για τόσα γίνονται εκεί. Και το θέμα δεν είναι μόνο πώς εμπλεκόμαστε στο πρόγραμμα εργασίας για το 2013, αλλά το τι ήδη έχει αρχίσει να προωθείται ε, για το 2014, 2020, στατικικό πρόγραμμα, πάρα πολύ σημαντικό λόγω της διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να κάνουμε όσον αφορά και το πρόγραμμα εργασίας ε, του, του ETF, του Ιδρύματος, αλλά γενικότερα τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που μια σε αυτή την δύσκολη περίοδο από πλευρά οικονομική, που θα είναι δύσκολη επομένω όχι μόνο για μα, αλλά θα είναι και για τι άλλε, για τι γειτονιάουσε χώρε. Έχουμε τώρα κάποιε τάσει ε, που έχουμε ξεχωρίσει και πρέπει να τις αναδείξουμε και παρακαλώ να τις προσέξετε. Είναι ότι όλο ένα και περισσότερο χρησιμοποιείται από πλευρά στρατηγικής ε, το Ίδρυμα. Το ανέφερε η Μαντλίν ε, ιδίω όσον αφορά τις ε, και ο συνάδελφο ο όσον αφορά τι χώρες της Βορειοαφρικής. Όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά σε όλη την Βόρεια Αφρική. Το 50% του πληθυσμού εκεί είναι κάτω από 25. Όμως είναι περιοχή υψηλού κινδύνου για πολλούς λόγους και το ότι επιστρατεύεται εκεί το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα και διεξάγεται διάλογος για κατάρτιση και επαγγελματικό προστατολισμό, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί και δεν αφορά μόνο το, το Ίδρυμα, αφορά την Ένωση γενικότερα. Εννοώ την ε, τάση για μία αηφόρο ανάπτυξη που προβλέπει στην της Λισαβόνας για να καταλάβουμε τι γνώσεις, τι δεξιότητες χρειάζονται. Ούτως ώστε να έχουμε όχι μόνο περιβαλλοντικό κεφάλαιο αλλά και ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο με κάποιο ευφύ τρόπο, ούτω ώστε να ανοίξουν τις εργασίες και επιχειρήσεις. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε τον ενδιαφέρον. Όχι μόνο δηλαδή να προσφέρουμε, αλλά να ελκύσουμε τον ενδιαφέρον. Να, τι χρειάζονται αυτέ οι χώρες που πολλέ από αυτέ έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και για αυτό το λόγο, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι κάτι σαν στρατηγική επένδυση. Πρόσφατα άκουσα ότι το Ίδρυμα έπρεπε να περικόψει το προσωπικό του 5% αλλά τώρα ε, πρόκειται να αυξήσει το προσωπικό κατά 2%. Αυτό είναι μια παραδοξότητα στις μέρες μας που έχουμε τόσο σημαντικές αλλαγές τώρα που έχουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Τι να σας πω, αυτό σαν, σαν φέτα σαλαμιού είναι. Σαλαμοποίηση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή σας να το εξετάσει καλύτερα, γιατί το να κόβονται οι πόροι, να απολύεται προσωπικό που ξέρει τη δουλειά, ακριβώς σε μια συγκυρία τόσο σημαντική και στρατηγική, ε, είναι όλο ένα πιο, πιο φανερό ότι έχουν προβλήματα, προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω το λόγο στους βουλευτές. Κύριε Θέρκας, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ειλικρινά να ευχαριστήσουμε τους τέσσερις διευθυντής και τους εμπειρογνώμονες. Και φυσικά να χαιρετήσουμε τον πρώην συνάδελφο Γιάννη Άντερσον. Μα τα είπαν οι διευθυντέ, μα τα είπαν οι εμπειρογνώμονε, μα είπαν το πώ λειτουργούν τα πράγματα. Μας, είπαν τι προβλέπεται για το μέλλον και νομίζω ότι αυτά τα οποία κάναμε αποτελεί παράδειγμα μίμηση και για άλλε υπηρεσίε. Σας ευχαριστούμε γιατί όλο αυτό το οποίο είπατε Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, σας ευχαριστώ. Τώρα που ξέρουμε ότι το ελεκτικό συνέδριο ήταν πάρα πολύ θετικό για το έργο σας. Εμείς το θεωρούμε αναμφίβολο. Και τέσσερις αυτοί οι οργανισμοί και υπηρεσίες. Θεωρούμε δεδομένο ότι επιτελούν πάρα πολύ σημαντικό έργο συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό ρεύμα. που χρειάζεται να έχει γερά θεμέλια στην πραγματικότητα αλλά και στην εμπειρογνωμοσύνη. Και άλλωστε όπως ξέρουμε μας έχουν βοηθήσει στο έργο μας πάρα πολύ αυτά τα ιδρύματα. Το Ρήνο και Μπιλμπάου. Είναι δύο ιδρύματα που καλέσαμε εδώ μέσω των προσώπων τους, ασχολούνται με πολύπλοκα ζητήματα, έχουν προβλήματα σημαντικά. Ας πούμε έχουμε το θέμα του, του, του κτηρίου στο Μπιλμπάου και θα πρέπει να δούμε μέσω της Ισπανικής κυβέρνησης τι θα γίνει με αυτή τη διεθνή συμφωνία. Και όπως έγινε στο παρελθόν θα πρέπει να δούμε πώς θα άρουμε αυτού του είδους τα διοικητικά προβλήματα. Λοιπόν, για πέστε μου για το μέλλον, τι θα κάνετε, τι θα γίνει, όχι το, το δικό σας, το δικό στρατηγικό πλάνο, τι γίνεται με το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο. Άλλωστε, στον ορίζοντα υπάρχουν πολλές απειλές για αυτό το αναντικατάστατο δικό σας το, το εργαλείο πολιτικής. Πρέπει να δούμε επομένως το θέμα το τόσο σημαντικό της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Και στο Τωρίνο είχατε να αντιμετωπίσετε ε, πολλά προβλήματα πρακτικά με το κτίριο κλπ. Για πέστε μας, είσαστε κοντά στο να βρείτε μια λύση. Επαναλαμβάνω, η σοσιαλιστική ομάδα ευχαριστεί. Και σας συγχαίρει γιατί το έργο το οποίο κάνετε επιτελείται με πολύ καλό τρόπο παρά τους περιορισμένους πόρους. Um, Έχοντας λοιπόν κατά νου το χρόνο, ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω πραγματικά να υποβάλλετε ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες. Επόμενος ομιλητής. Εγώ θα σας απογοητεύσω, δεν θα υποβάλω ακριβώς ερώτηση, αλλά ήθελα να πω ότι πραγματικά αξίζουν τον κόπο τα λεπτά που δίνουμε σε αυτές τις επιτροπές. Επίσης, ε, θέλω να σας πω ότι τα στατιστικά δεδομένα μιλάνε από μόνο τους. Έγινε αρκετός λόγος για την δουλειά αυτών των Ιδρυμάτων. Γνωρίζω από τις επισκέψεις μου στο Μπιλμπάο και από την σχετική στο σελίδα ότι οι υπηρεσίες τους είναι ε, πολύτιμες. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που πήγα στο Σεντεφόπ. Θέλω όμως να πω κάτι ε, σχετικά με αυτό που είπε ε, ο Γιάνν Άντερσεν και για το Τουρίνο. Ο Γιάνν είπε ότι χρειαζόμαστε ε, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και συνέπεια. Έτσι λοιπόν με τις περικοπές υπάρχουν προβλήματα επάντρωσης και ίσως το ίδιο να ισχύει και για άλλους ε, φορείς. Ε, η δική μας ευθύνη και της Επιτροπής Προεπολογισμών, αλλά η δική μας κυρίως είναι να δείξουμε στην Επιτροπή Προεπολογισμών ότι πρέπει να κάνει πολιτική αξιολόγηση και όχι οριζόντιες περικοπές σε όλα τα ιδρύματα. Γιατί υπάρχει μια τάση στην Επιτροπή Προεπολογισμών να αντιμετωπίζονται όλα τα ιδρύματα ε, με τον ίδιο τρόπο, οριζόντιες όπως σας είπα ε, περικοπές, να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι αυτό που είπα ε, θα ληφθεί υπόψη στον προπολογισμό ε, που θα συσταθεί κατά το τέλος του έτους. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω ε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις ο καθένας για δύο λεπτά. Zlato check, please. Thank you. I would like to start uh, uh, the questions related to... Κύριε Στάτλατσεκ, για το θέμα του Μπιλμπάου, να πω ότι καταφέραμε να έχουμε, αν μη τι άλλο, ένα βασικό κείμενο για την συμφωνία περί έδρας. Με την Ισπανική κυβέρνηση φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, θα υπογραφεί, αλλά χρειάζεται χρόνο διαδικασία για τα περισσότερα υπουργεία. Πρέπει να υπογράψουν τις διεθνείς συμφωνίες, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας. Η δυσκολία είναι να πάρουμε την υπογραφή για τη συμφωνία της έδρας με θέματα όπως τις ασφαλίες των κτηρίων, την πρόσβαση στη δημόσια υγεία και βεβαίως να υλοποιηθούν και τα σχετικά μέτρα όπως αναφέρονται στην συμφωνία. Μιλάμε εδώ για τη χώρα των Βάσκων. Μετά τι υπογραφέ τη κεντρική κυβέρνηση, θα πρέπει να έχουμε διαπραγματεύσει με την ίδια τη χώρα των Βάσκων, την περιφερειακή δηλαδή και κυβέρνηση, και να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα μέτρα που ε, αναφέρονται. Για την ώρα το κτίριο δεν έχει περιληφθεί στη Συμφωνία ε, Έδρας, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η κρίση. Πάντως, ε, στον οργανισμό καταφέραμε να αρχίσουμε μια έρευνα αγοράς για να αναζητήσουμε το κατάλληλο κτίριο και αυτό σκοπό έχει να ικανοποιήσουμε και το αίτημα για περιορισμό των ε, δαπανών στους περισσότερους τίτλους. Ίσως να βρούμε χαμηλότερο ενίκιο επιμίσθιο και να έχουμε ένα άλλο κτίριο με καλύτερες συνθήκες εργασίας, Διότι κάποιοι από εσάς μας επισκεφτήκατε στον Μπιλμπάου και ξέρετε ότι η οργάνωση για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εργάζεται σε συνθήκες που δεν είναι και καλύτερες. Ουδέποτε προβλέφθηκε το κατάλληλο κτίριο για τα γραφεία τους. Οπότε, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε χαμηλότερο επιμίσθιο αλλά και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Εάν θέλετε τη στήριξή μας, μάλλον εάν μιλάτε για στήριξη, καλοδεχούμενη κάθε είδους στήριξη, ειδικά από βουλευτές και μάλιστα της Ισπανίας. Ξέρω ότι η κυβέρνηση της χώρας των Βάσκων χαίρεται που βρισκόμαστε εκεί. Γιατί και άλλε συνδικαλιστικές οργανώσει και άλλοι εταίροι θέλουν να είναι σε, συνεργασία, σε στενή συνεργασία μαζί μα. Η Βάσκη, λοιπόν, η περιφερειακή κυβέρνηση, θα μας στηρίξει στον οργανισμό για την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας. Στην Ισπανία, ακριβώς σε επίπεδο εταιρεών υπάρχουν πολλές δυσκολίες προκειμένου να σεβαστούν τις προσδιαγραφές. Να είναι υψηλό το επίπεδο της ε, καλής ε, εργασιακής υγείας. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε στενότερες επαφές μαζί τους για να τους υποστηρίζουμε. Τώρα, Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Αλλά με συγχωρείτε, πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Κύριε Λετμαγερ. Δεν μου απευθύνθηκε συγκεκριμένη ερώτηση, οπότε θα είμαι ιδιαίτερα σύντομα. Σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα στη διαδικασία του προπολογισμού. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να είναι εύληπτα όλα αυτά και να σα παρουσιάσουμε τα κατάλληλα επιχειρήματα. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να λάβουμε τα κονδύλια τα οποία ζητούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μενέντες Βάλδες. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Πολύ πολύ σύντομα. Θέσατε ερώτημα για το εάν έχουν διοριστεί προγνωμόνε από το Κοινοβούλιο. Όχι νομίζω. Όπω και ο κύριο Λεπμάγερ. Βρισκόμαστε στην ίδια θέση με τη ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Είμαστε από του παλιότερου οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λόγω τη κοινων... κοινή προσέγγιση που υιοθετήσαν τα θεσμικά όργανα, ίσω ίσως στο μέλλον να υπάρξουν προτάσει για την αναθεώρηση του ιδιωτικού μα κανονισμού βάσει τη συνήθου νομοθετική διαδικασία. Πολύ σύντομα να απαντήσω και για τι μειώσει των κονδυλίων και το προσωπικό. Ναι, κάποιε εξοικονομήσει μπορούμε να κάνουμε, αλλά αγωνιζόμαστε να το πετύχουμε. Είμαστε σχετικά μικρός φορέας. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Εάν κόψετε ένα σημαντικό κονδύλι, αυτό θα σημαίνει περισσότερο μείωση δραστηριοτήτων. Έχουμε 20 εκατομμύρια προπολογισμό με μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων εσωτερικές, μέρος της έρευνας εντός οργανισμού. Για το λειτουργικό αυτό προπολογισμό έχουμε 8 εκατομμύρια και μία από τις τρεις μελέτες που καλύπτουμε αφορά 32 χώρες, κράτη-μέλη και υποψήφιες χώρες και δίνει κέρδος 3 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το ποσό. Εάν πρέπει να εξοικονομήσουμε ποσά, κονδύλια, θα πρέπει να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις από τους πολιτικούς ηθήνοντες και από εμά. Ας το έχουν υπόψη τους λοιπόν οι υπεύθυνοι θα μειωθεί το επίπεδο και όγκο των πληροφοριών που μπορούμε να παράσχουμε από τον οργανισμό μας. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας στην Επιτροπή Απασχόλησης. γιατί εκτός από εσάς μας στηρίζουν και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, μας, καταφέ, μας επιτρέπουν να έχουμε στρατηγικότερη προσέγγιση, πιο ε, σκόπιμη στις περισσότερες χώρες παρέμβασής μας. Να απαντήσω στην ερώτηση για το κτίριό μας. Από την ε, στιγμή της επίσκεψής σας, λίγα έχουν γίνει. Είμαστε κοντά στο να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα στα τέλη της περσινής χρονιάς αλλά μετά από απόφαση της κυβέρνησης να μην συνεχίσει τις ε, διαπραγματεύσεις λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Ιταλία, έχουμε βρεθεί πάλι στο μηδέν στην αρχή. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εκλογών 24 και 25 Φεβρουαρίου για να δούμε ποιος θα αναλάβει και ποιος θα είναι ο συνομιλητής μας για να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν αρκεί να έχουμε συμφωνία για την έδρα. Τέτοια συμφωνία υπάρχει. Επικαιροποιήθηκε το 2012 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο, αλλά το πρόβλημα είναι η εφαρμογή της. Ως προς την επιλογή του κτηρίου δεν έχει επιτελεστεί πρόεδρος. Αλλά να σας καθησυχάσω. Μαζί με το ελεγκτικό συνέδριο που μας επισκέφτηκε επανειλημμένος, το τόνισαν αυτό και στην έκθεσή του, στη δεύτερη εκδοχή της που θα σας δοθεί σύντομα, τον οργανισμό μας κοιτάζουμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας. Οπότε έχουμε μια σύμβαση προσωρινή για ένα χρόνο με ε, εξωτερικούς νομικούς συμβούλους και κοιτάζουμε κατά πόσο μπορούμε να προσφύγουμε για να διεκδικήσουμε τα νομικά μας δικαιώματα και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας σε αυτό το θέμα η διπλωματική οδός έχει και τα όρια της. Τώρα μπορεί να χρειαστεί να αναλάβουμε δράση για να μετακινήσουμε την έδρα μας καπαλού ως προς την στήριξή σας. και τη διαφοροποιημένη προσέγγιση προς τους διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να έχουν υπόψη ότι ό,τι επιτυγχάνουμε έχει να κάνει με 2,5% ε, προσωπικό επάντρωση αναχώρα. Αλλά με τέτοια επάντρωση δεν μπορεί κανείς να επηρεάσει την ε, κατάσταση και την εξέλιξη των ανθρωπίνων πόρων στην κάθε χώρα. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ που μας ε, στηρίξατε την Επιτροπή Βασχόλης και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι βρεθήκατε. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι βρεθήκατε εδώ. Πάμε λοιπόν στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Η Ιούτα Στάινοχουκ είναι η συγγήτρια και σήμερα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για τις 21 ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι εξαγορές ε, επιχειρήσεων ε, είναι κατ' ουσίαν βοηθητικές, βοηθούν την οικονομία να παραμείνει ανθυρή και επίσης ε, να λειτουργούν καλύτερα επιχειρήσεις. Αλλά εμείς ε, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά και επίσης να ε, θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμβάλλουν στο να διατηρούνται θέσεις εργασίας ε, στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν στο δικό μου το σχέδιο έκθεση σε ιδιαίτερη σημασία αποδίδω σε αυτό που είναι σημαντικό για την Επιτροπή Επασχόλησης, δηλαδή στην κατάσταση των εργαζομένων ε, στις εκπροσωπήσεις των εργαζομένων, ε, στα δικαιώματα των απασχολούμενων, στη συναπόφαση. Συνολικά λοιπόν έχουμε 21 ε, τροπολογίες τις οποίες έχουν καταθέσει το ΕΛΚ και η ΑΛΔΕ. Και από ό,τι φαίνεται οι συντηρητικοί συνάδελφοι σε θέματα εργαζομένων και συνδικάτων ε, κρίνουν ότι προχώρησα πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι στις ε, συμβαστικές προτάσεις θα μπορέσουμε κάπως ε, να τα βρούμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν ορισμένα θέματα όπου πρέπει να συζητήσουμε λιγάκι. Στις τροπολογίες 12 και 16 Πρόκειται για τις εκπροσωπήσεις των ε, εργαζομένων μιας επιχείρησης. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι ε, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα ανεξάρτητα συνδικάτα. Στην Ευρώπη ε, το τοπίο των συνδικάτων ποικίλει πάρα πολύ και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτούς το στις υπόλοιπες τροπολογίες πρόκειται για τη διατήρηση των συνδικάτων κατά τη διάρκεια της εξαγοράς. Νομίζω όμως ότι έχουμε συζητήσει και σε άλλες ε, εισηγήσει όπου έχει καταστεί απόλυτα σαφές ότι πριν από την εξαγορά οι, ε, τα συνδικάτα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Στην τροπολογία υπερθμών 15 πρόκειται για το κόστος ε, που προκαλείται από ε, την πρόσληψη ειδικών. Εγώ πιστεύω ότι ε, τα συνδικάτα δεν μπορούν ε, να πληρώνουν κάτι τέτοιο από τις εισφορές των μελών. Νομίζω εδώ πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι ίδιες επιχειρήσεις οφείλουν να καλύπτουν αυτό το κόστος. τώρα είμαι σε φάση όπου επεξεργάζομαι τις συμβαστικές προτάσεις, ε, θα τις καταθέσω μέχρι το τέλος εβδομάδας στους σκιώδεις εισηγητές και την επόμενη εβδομάδα ε, θα συναντηθούμε οι σκιώδεις εισηγητές ε, για μια περιττέρω συνάντηση. Νομίζω ότι τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό έτσι ώστε να στηρίξουμε όλη αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν μιλώ ως ε, συντονιστής, αλλά ως ε, σκιώδης εισηγητής. Αναμφίβολα ότι όταν έχουμε αναδιάρθρωση, εξαγορά, ε, ας πούμε κάποιες εταιρείες ότι θα πρέπει να καλύπτουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Και επίσης είναι συνεχής ο αγώνας του πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και τι θα κάνουμε. Ότι μπορούμε τόσο να μπορούμε να δώσουμε μια όθηση σε αυτή την καινούργια κατάσταση της οικονομίας, πώς θα βρούμε μια ανάπτυξη, πώς θα έχουμε ευελιξία, πώς θα έχουμε ασφάλεια ταυτόχρονα. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε το ότι είναι πάρα πολύ βασικό το πώς θα βρεθεί η μέση οδός. Πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να καλύψουν και να εξισορροπήσουν τα συμφέροντα και της εταιρείας αλλά και των εργαζομένων. Όσον αφορά τώρα το κείμενο το οποίο τώρα μελετούμε, υπάρχει κάποια έλλειψη ισορροπίας. Ε, πολλές φορές έχουμε κάποιες επαναλήψεις βέβαια, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά αυτές τις επαναλήψεις μπορούμε να επαναδιατυπώσουμε κάποιες διατάξεις, κάποιου είδου ε, παραγράφους, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που νομίζω επίσης ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες διαγραφές, κάποιες απαλήψεις κάπου στη διάταξη 9 νομίζω γράφει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όσο, όσο δεν έχουν δώσει το πράσινο φως οι μισθωτοί Δεν είναι ορθό αυτό. Δεν στέκει αυτό. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Επίσης, η χρηματοδότηση θα γίνει με κάποιο είδους ε, χρηματοδότηση της επιχείρησης, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε στους εκπροσώπους εργαζομένων, δεν μπορούμε να τους δώσουμε το δικαίωμα του βέτο ε, για αυτές τις διαμετρήσεις, γιατί αυτό ε, ενδεχομένω έχει, έχει αρνητικό αποτέλεσμα και σε επιπτώσεις, διότι αν έχουμε ας πούμε ένα συνδικάτο το οποίο είναι πάρα πολύ πεισματικό, τότε αυτοί αν είναι αρκετά σκληροί. Αν, επιμείνουν πολύ, τότε ίσως οδηγήσουν στην ε, ματέωση μιας εξαγοράς ή ακόμα και στη χρεοκοπία της ε, επιχείρησης, εάν μπλοκαριστεί η εξαγορά. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε περισσότερη ε, περισσότερη εξισορροπή Νομίζω ότι το 13 υπερβάλλει κάπως. Για να δούμε. Τι δυνατότητε πάνε σε Ευρώπη. Για να δούμε τι αρμόδιε έχουν τα κρατη σε σχέση με αυτό. Εγώ πάντω με μεγάλη μου χαρά μπορώ να συνεργαστώ ε, με την επεξεργασία, με τη διεκπαιρέωση αυτή τη έκθεση. Καλωσορίζω τις δηλώσεις ε, της εισηγήτριας ότι είναι πρόθυμοι να αναζητήσουμε συμβαστικέ λύσει. Σε κάποιε περιπτώσει όντω θα έχουμε κάποιε δυσκολίε, διότι όντω υπάρχει απόκληση απόψεων. Σοβαρέ αποκλήσει, περίπου στι γραμμέ αυτό που περιέγραψε ο κ. Όρη. Σε συνθήκε κρίση, οι εξαγορέ θα λάβουν χώρα σε πολλέ περιπτώσει με σκοπό τη διάσωση επειδή είναι έκτακτες οι περιστάσεις. Ενώ σε πιο συνηθισμένες ε, καταστάσεις ο σκοπός είναι ο αντίστροφος. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις εταιρείες να αναδιαρθρωθούν και καλά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ε, προωθήσει το θέμα αυτό για την ερχόμενη πενταετία. Να βασιστεί σε εταιρικέ συμφωνίε για να προστατεύονται και οι εργαζόμενοι σε διάφορε εταιρείε. Και για εταιρείε ιδίω που έχουν λάβει ορθέ αποφάσει για να παραμείνουν ε, στην αγορά. Πέραν των επιφυλάξεών μου βέβαια, προσπάθησα να είμαι επικοδομητικό στι ε, τροπολογίε μου, όμω κάπω προκαλεί σύγχυση η πρόταση ότι οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν ευθύνη έναντι των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εταίρων εφόσον υπάρξει προσφυγή σε πρωτοδικείο. Αλλά αυτό είναι πρωτογενή λειτουργία των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων, όχι των εργοδοτών. Επίση, οι εξαγορέ θα πρέπει να εγκρίνονται από συμφωνίε των κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι συζητήσιμο. Και πέραν αυτού, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι εξαγορές θα πρέπει να αναστέλλονται εφόσον υπάρχει έστω και μία αντίρρηση ή έστω και μία διαρκής ε, προσφυγή παράπονο. Αυτό δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό, διότι σωρευτικά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να μείνουν όλοι άνεργοι γιατί μια εξαγορά παρεμποδίζεται. Έχουμε υποβάρει λοιπόν τροπολογίες που θα πηχήσουν τις ε, επιφυλάξει μα και ευχαριστώ να ακούσω τι παρατηρήσει και των συναδέλφων. Ελπίζω να βρούμε κάποιο πεδίο συνεννόηση, αλλά με ενθαρρύνει σε κάθε περίπτωση η αρχική τοποθέτηση τη εισηγήτρια που δήλωσε πνεύμα ευελιξία. Uh, ευχαριστώ να δώσω πάλι το λόγο στην εισηγήτρια. Yeah. Ευχαριστώ πολύ τους ε, συναδέλφους ε, για όλα αυτά που είπαν. Νομίζω ότι την επόμενη ε, Δευτέρα θα συζητήσουμε για τις συμβαστικές προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί. Και θέλω να σκεφτείτε το εξής, ότι και τα συνδικάτα ενδιαφέρονται να έχουν μια καλά λειτουργούσα επιχείρηση κυρίως όταν τίθεται θέμα εξαγοράς. Γιατί και τα συνδικάτα δεν ενδιαφέρονται, δεν θέλουν να καταστρέφουν θέσεις εργασίας. Το αντίθετο θα έλεγα. Αν δει κανεί λιγάκι το ευρωπαϊκό τοπίο, διαπιστώνει ότι η συμπερίληψη των ε, συνδικάτων σε οικονομικές ε, αποφάσεις είναι πιο σημαντική στις χώρες ε, που και οικονομικά είναι πολύ ισχυρές. Πολύ ωραία. Ε, στις 21 Φεβρουαρίου θα ε, υιοθετηθεί η έκθεση. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο 17. Η κινητικότητα των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ Έχουμε εισηγητή ε, τον κύριο Σόγκορ. Ε, πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο της αμέσως στον εισηγητή. Ε, θα μιλήσω ουγγρικά következő javaslatokat fogalmaztuk meg eh, ebben a véleménytervezetben. Egy fok... Να σας πω κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες στην Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ιών. Να δούμε πώς Πώ θα σταματήσει η εκμετάλλευση των γυναικών. Τρίτον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν να υπάρχει περισσότερη ε, καταπολέμηση ε, του δουλεμπορίου και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα σεβαστούμε την πολιτιστική ε, διάσταση, παράδοση, κυρίως όσον αφορά τις, τις μειονότητες και να δούμε με ποιο τρόπο θα προστατευτούν τα δικαιώματα των γυναικών. Πώς τι θα γίνει τα εθνικά προγράμματα της ε, αναδιάρθρωσης. Επίσης λέμε ότι θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα οριζόντια και εξειδικευμένη για, για τις καλές πρακτικές και, και να έχουμε αποτελέσματα σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο και επίσης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τα προγράμματα εθνικά κλπ. ούτως ώστε να εμπλακούν οι γυναίκες σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και την κοινότητα και επίσης θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να διευκολύνουν τις διαδικασίες για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και έτσι να έχουμε αυτό το, το αίσθημα του ανήκειν στην κάθε κοινότητα. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τις συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών στις, ε, στις κοινότητες αυτές των, των εκπατρεσμένων. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις, ε, τις διαδικασίες κοινωνικής ε, ένταξης, της παροχής ψυχολογικών ε, συμβουλών για την κατανόηση των προβλημάτων. Να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επίσης, κάποιο είδου ε, υπηρεσιών παροχή συμβουλών για να μπορούν να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό και στην εργασία γυναίκες. Επίσης είναι σημαντικό ε, να καταλάβουμε τις, ε, τις συνήθειες ε, στις χώρες που πάνε να κατοικήσουν οι γυναίκες. Επίσης θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την αμοιβή αναγνώριση των τίτλων σπουδών, διπλωμάτων και θα πρέπει να γίνεται γρήγορα αυτή η διαδικασία της αναγνώρισης των ε, τρίτων σπουδών. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην κυρία Μπλινκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτο, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, γνωμοδότηση αυτή γιατί τα περισσότερα σημεία που αναφέρατε είναι σημεία που θα υποστηρίξω. Λόγω της σημερινής κατάστασης, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε να αυξάνεται η κινητικότητα των γυναικών. Πολλά προβλήματα σχετίζονται με αυτό το φαινόμενο. Θα ήθελα να θίξω κάποια σημαντικά στοιχεία χέρι με χέρι με τους ε, εισηγητές σκιώδη και μη, θα προσπαθήσουμε να εξέφερουμε τις καταλληλότερες λύσεις. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικεντρωθούμε στην υγεία των γυναικών, την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που γνωρίζουν κάποιες γυναίκες, όταν ε, μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και για, τον, για, τη, για το χάσμα, το μισθολογικό που παραμένει χωρίς να βρίσκονται οι άντρες και οι γυναίκες στο ίδιο επίπεδο. Θα πρέπει επίσης οι γυναίκες να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ε, Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ηλικιακές ομάδες, διότι τα προβλήματα των νέων γυναικών και των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών μπορεί να διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Λόγω της κατάστασής τους, της θέσης τους και των ευκαιριών που τους προσφέρονται. Θα έλεγα στη γνωμοδότηση να δοθεί έμφαση τη διάσταση που αφορά τα επαγγελματικά προσόντα των γυναικών. Αυτά όμως που έχουν κατακτήσει λόγω της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Η διάσταση της διαβίου μάθησης και της εκπαίδευσης ή κατάρτισης πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία ώστε οι γυναίκες να βρουν μια θέση εργασίας ώστε να μπορούν να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Επίσης, πρέπει να δούμε το συσχετισμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Τη δυνατότητα των γυναικών να διαχειρίζονται τον χρόνο τους, χρόνο εργασίας και ελεύθερο, και αυτό εφόσον μιλάμε για πλήρη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πτυχές, αλλά νομίζω ότι θα τις καλύψω όταν ξανασυζητήσουμε τη γνωμοδότηση αυτή ή στι διμερεί μα δοθές. Προεδρο, ευχαριστούμε. Ας ξανακούσουμε τον εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν το συμπεριέλαβα στην έκθεση. Ελπίζω όμως Ελπίζω ότι οι κυρίες θα το σημειώσουν αυτό. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια έκθεση που συντάσσει άνδρας απευθυνόμενη προς τις γυναίκες και προβλήματα γυναικών. Πρόεδρος, ευχαριστώ για τις εφαρμογές της ψηφιακής υπογραφής. Θα γίνει μια δοκιμή με την έκθεση αυτή. Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοια δοκιμή στις 18.45. για την υποβολή τροπολογιών 31 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Εξέταση τροπολογιών 21 Φεβρουαρίου. Συμβαστικές τροπολογίες 20 Μαρτίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Επασχόλησης 21 Μαρτίου και Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2013. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν ε, στο σημείο υπερθμών 18 της σημερινής διάταξης. Ε, πρόκειται για την ε, προστασία επεξεργασίας δεδομένων. Εδώ είμαι εγώ η εισηγήτρια και σήμερα θα εξετάσουμε και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Λοιπόν, μου δίνω το λόγο και ευχαριστώ τους εισηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ε, είχαμε μία σύντομη ε, συνάντηση για να καθορίσουμε και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε επειδή εγώ την έκθεση κατ' ουσίαν την περιόρισα στο άρθρο 82 ε, και θέλησα να δώσω κυρία ιδιαίτερη έμφαση στην Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων. Ε, εκατόν τόσες ε, τροπολογίες κατατέθηκαν, προέκυψαν διάφορα θέματα από αυτές τις τροπολογίες και θα αναφερθώ σε αυτά τα θέματα. Ένα θέμα είναι η μαύρη κατάλογη, δηλαδή η κατάλογη αυτή έτσι ώστε εργαζόμενοι που ε, συνδικαλίζονται να καταγράφονται σε αυτούς τους καταλόγους. Πήραμε τροπολογίες ε, για το θέμα αυτό και ε, θα προσπαθήσουμε να καταθέσουμε, να συντάξουμε συμβαστική πρόταση. Το δεύτερο θέμα αφορά την εθελοντική συμμετοχή, κατά πόσον ισχύει αυτό ή όχι. Πρόκειται για το άρθρο 7 ε, ε, για το σημείο 7 της πρώτης κομισιόν. Το τρίτο μπλοκ αφορά ε, τον ίδιο τον εντεταλμένο για την προστασία δεδομένων, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν και για αυτόν δεδομένα και προστασία δεδομένων για αυτόν συγκεκριμένα και πώς θα γίνεται όλο αυτό. Κατόπιν, ένα άλλο θέμα είναι κατά πόσον θα πρέπει να καθορίζεται ε, αν θα λαμβάνεται υπόψη η, ο αριθμός των ε, συνεργατών σε σχέση με τον εντεταλμένο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά ε, την ενημέρωση μέσα στο εσωτερικό της επιχείρησης τόσο όσον αφορά το άρθρο όσο και το, αιτιολογώντας ε, το ε, εδάφιο 124 του αιτιολογικού. Πάρα πολλές ε, τροπολογίες αφορούν στις κατεξιδότηση πράξης και εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, ποικίλουν δηλαδή του χρόνου, με συγχωρείτε, την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Κατατέθηκαν και πολλά άλλα θέματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν θα σας τα αναφέρω λεπτομερώς. Ίσως εδώ οι σκιώδεις συζητητές επιθυμούν οι ίδιοι να αναφέρουν τι είναι σημαντικό για αυτούς, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης. Αυτά είχα εγώ καταρχήν να σας πω. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο τους συναδέλφους ε, και πρώτα απ' όλα στην κυρία Ρέγνερ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και η συγκήτρια. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Η προστασία των δεδομένων είναι πραγματικά ένα θέμα που αφορά όλους τους απασχολούμενους και θα έπρεπε να είναι γεμάτη η αίθουσα και πολύ ζωντανή συζήτηση αλλά επειδή είναι περασμένη ώρα εγώ θα είμαι σύντομη και θέλω να πω ότι η δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα ε, σε συνεργασία με τους σκιώδης ηγητές είναι πάρα πολύ επικοδομητική και πραγματικά είναι χαρά για μας να συνεργαζόμαστε μαζί σας. Ε, οι τροπολογίες ε, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, υπάρχουν αρκετά που αξίζουν τον κόπο να εξεταστούν. Εγώ σύντομα θα αναφερθώ σε τρία θέματα. Το πρώτο θέμα είναι ο εντεταλμένος για την προστασία των δεδομένων. Αυτός είναι ο άνθρωπος κλειδί για τους απασχολούμενους, για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί του ε, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία δύο κατηγοριών ε, επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει τέτοιος εντεταλμένος ή αρμόδιος και άλλες επιχειρήσεις όπου να υπάρχει. Είναι πολύ σημαντική η προστασία των δεδομένων και είναι και σημαντικό να έχουμε κατά νου αυτός ο άνθρωπος να μην ε, τα έχει πιάξει πλακάκι αν θέλετε πολύ απλά με την επιχείρηση. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός πρέπει να έχει μια ισχυρή θέση ε, να προστατεύει τους εργαζόμενους από καταγγελίες συμβάσεων και παρεμφερεί. Ε, το άλλο, οι μαύροι κατάλογοι, ε, blacklist όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι έχουμε δει ότι επανεμφανίζονται τη οι μαύροι κατάλογοι. Οι μάλιστα τις ε, ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα της Επιτροπής μας να είναι σαφές ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις ε, και αυτές, ε, αυτοί οι μαύροι κατάλογοι είναι καταδικαστέοι. Μόνο απευθυντική θηρίδα αυτή η αρχή. Για ποιον να ισχύει one stop shop. η εργαζόμενοι που ε, εργάζονται στην Google ας πούμε έχουν πρόβλημα και πού θα πρέπει να απευθυντούν αυτή η αρχή της μοναπευθυντικής ε, θηρίδας μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα στους εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι εργαζόμενοι ε, εάν υπάρχει θηγατρικοί να μπορούν να απευθυνθούν στο δικό τους ε, τον διεταλμένο που είναι στη χώρα τους. Γιατί όσο πιο μακριά είναι επιχείρηση, τόσο πιο πολύ δυσκολεύει η κατάσταση. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα πάρα πολλούς τομείς όπου απλά η γεωγραφική απόσταση και η απόσταση γενικότερα δημιουργούν ε, πρόβλημα στους εργαζόμενους ε, στο να απευθυντούν στον ε, εντεταλμένο για την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρέπει να ευχαριστώ και εγώ όλους όσοι κατέθεσαν τροπολογίες. Για λόγους αρχής θέλω να πω ευθύς εξ αρχής ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης η προστασία των δεδομένων πρέπει να παραμένει πιστή στις διατάξεις του άρθρου 82 του κανονισμού. Βεβαίως κατανοώ πολύ καλά ότι η προστασία δεδομένων μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις και ιδέες, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παραμένουμε στις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής. Εγώ πιστεύω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η προστασία των δεδομένων ε, πρέπει να καθορίσει ελάχιστες προδιαγραφές, γιατί κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στους εθνικούς νομοθέτες να προβλέψουν εξαιρέσεις από αυτόν τον κανονισμό. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πρέπει να πω η τροπολογία 82 του Jean Lambert προβλέπει ε, κατά την άποψή μου ε, μια καλή περιγραφή των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την έκθεση. Όσο αφορά το άρθρο 82 παράγραφος 1 του κανονισμού, διαπίστωσα ότι αρκετές ε, τροπολογίες είναι περίπου ίδιες στο περιεχόμενο. 83, 84 και 85 παραδείγματος χάρη. Και αυτό δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί συνένεση. Βέβαια, αυτές οι τροπολογίες ενέχουν και το ίδιο λάθος. Δηλαδή επαναλαμβάνουν ε, τον όρο ε, συλλογικές συμβάσεις. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι τυπογραφικό λάθος. Ε, το 82 στον κανονισμό, εκεί διαπίστωσα ότι αρκετές τροπολογίες που αφορούν στους μαύρους καταλόγους, ένα θέμα που έχουμε εξετάσει παλαιότερα, στην έκθεση Ντελή για την υγεία και την ασφάλεια. Εκεί ε, υπάρχουν αυτές οι τροπολογίες. Το θέμα λοιπόν είναι πολύ ευαίσθητο και ορισμένες από τις ε, τροπολογίες αυτής της έκθεσης ε, επικαλούνται κυρώσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επειδή υπάρχουν όλα αυτά, πρέπει να γίνουν ε, περισσότερες συζητήσεις. Άρα δηλαδή πρέπει να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε με την πρόταση για κυρώσει σε εθνικό επίπεδο. Οι 92, 93, 94, 95 και 100 αυτές οι τροπολογίες μοιάζουν. Και βεβαίως συμφωνώ ότι ε, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους ως ε, στοιχείο ε, διακριτικής μεταχείρισης. Θα πρέπει να προστατεύεται πάντα η ιδιωτική σφαίρα. Βέβαια, νομίζω ότι η τροπολογία υπαριθμών 95 ε, μπορεί να συζητηθεί γιατί αναφέρει και παραθέτω ένας ε, επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, δεδομένα για την σεξουαλική ζωή, τις πολιτικές πεπιθήσεις, τις θρησκευτικές πεπιθήσεις και το ποινικό μητρό του εργαζόμενου. Το κατανοώ αυτό, αλλά εννοεί αυτή η τροπολογία ότι ένας εργοδότης δεν μπορεί να ζητήσει ποινικό μητρό αν έχει λευκό ποινικό μητρό ένας εργαζόμενος. Αυτό δεν είναι λογικό. Ξέρετε ότι εδώ ας πούμε για να προσληφθεί κάποιος ε, πριν υπογράψει πρέπει να ε, καταθέσει ε, στοιχεία για το λευκό ποινικό του μητρό Και η τροπολογία 96 λέει ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να ελέγχουν τη δουλειά του εργαζόμενου. Αν το κάνουμε όμως αυτό στις επιχειρήσεις, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα για τις οικονομίες μας. Ε, διαφωνώ επίσης ε, με την τροπολογία υπαριθμών 118. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι εθνικές νομοθεσίες επικύλουν όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων. Και επανέρχομαι σε αυτά που είχα πει στην αρχή, ότι η έκθεση αυτή πρέπει να έχει κατά νου ελάχιστες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι ε, μια άκαμπτη πανευρωπαϊκή νομοθεσία. Και πιστεύω, παρά τις αντιρρήσεις μου, ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση για συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί ένας καλός συμβασμός. Σας ευχαριστώ και συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μας αφορούν πολλούς, ξημών τέλο πάντων και είναι θέμα του να προσπαθήσουμε να βρούμε την ακριβή διατύπωση η οποία θα ταιριάζει με διάφορες τροπολογίες. Αυτό που μας είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά και μία από τις σκέψεις που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το πώς όλα αυτά θα συναρμόσουν το ένα με το άλλο μέσα στον κανονισμό και πώς θα είμαστε σαφέστεροι. Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο παντού. Έχετε δίκιο στην ανάλυση σας για τα θέματα σε σχέση με το μέγεθος της εταιρείας, τη υπηρεσία προστασίας δεδομένων, την δικαιοδοσία αρμοδιότητα. Για πρέπει να δούμε και την γεωγραφική διάσταση. Μπορούμε όλα αυτά πάντως να τα συνδυάσουμε στις προτάσεις μας. Τώρα το θέμα είναι ο σκοπός της συλλογής δεδομένων. Να μπορεί κανείς να έχει ό,τι χρειάζεται σε σχέση με τα προαπαιτούμενα του νόμου. Σε σχέση με τους τρίτους, σε σχέση με τα κοινωνικά επιδόματα, δεν μπορούμε όλα αυτά να τα αποκλείσουμε γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία σημαντικά τα οποία δεν χρειάζεται κάποιος εργοδότης. Α πούμε να ξέρει τα σχετικά με τη μητρότητα, ε, την ασθένεια, την υγεία κλπ. Τώρα για το ποινικό μητρό υπάρχει εδώ ένα ζήτημα σε σχέση με το εάν κανείς δεν μπορεί να ψάξει το ποινικό μητρό, Τι θα γίνει με κάποιους ε, που έχουν ε, διαπράξει εγκλήματα σε σχέση με τη γενετήσια ζωή. Δηλαδή έχουμε ε, και κάποιους που έχουν διαπράξει παιδική πορνογραφία κλπ. κλπ. Θα πρέπει και αυτό να δούμε με συνέπεια πώς θα το καλύψουμε. Επίσης θα πρέπει να είμαστε και σαφείς. Για ποιο λόγο ζητείτε αυτή η πληροφορία. Να μην είμαστε παράλογοι, ούτε κανείς να μην μπορεί να βρει δουλειά. Ανάλογα βέβαια με το τι ποινική καταδίκη έχει υποστεί. Έχουμε τώρα όλα αυτά τα στοιχεία και άρα θα πρέπει να δούμε πόσο ευρεία θα να είναι η ρύθμιση. Έχουμε δύο ή τρία άρθρα που το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο στον αφορά την ατολική γιατί έχουμε κάποιες ε, ε, Προβλέψει οι οποίε όντω καλύπτουν τις ανάγκες της απασχόλησης. Υπάρχουν και κάποια ε, σε άλλε τροπολογίες που από την δική μου ε, πολιτική ομάδα γιατί ακριβώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ από τη δική μου πολιτική ομάδα η συγκεκριά. Οπότε προσπαθούμε να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα και εσωτερικά. Να δούμε τι θα γίνει από πλευρά απασχόληση λοιπόν. και θα υποβάλουμε τροπολογίες όπου χρειάζεται. Gut, dann ähm, erst einmal herzlichen Dank für die Rückmeldung. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Νομίζω λοιπόν ότι ακριβώς αυτό ε, θα κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις ε, τροπολογίες σε συμβαστικές ε, προτάσεις και βεβαίως ε, δεν θέλουμε να υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές ε, και θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Και τις ε, συμβαστικές προτάσεις θα τις συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας στις 20 Φεβρουαρίου και στις 21 θα ψηφίσουμε. Και πάμε στο τελευταίο σημείο της μερίσιας διάταξης, στο 20. Που αναβλήθηκε για την επόμενη φορά και το 21. Και το 21 επίσης αναβάλλεται για την επόμενη φορά. Ο συγητής, ο κύριος Μπουλόν, δεν είναι εδώ, ούτε και η σκιώδη συγήτρια Κατόπιν τούτου ε, την επόμενη φορά θα εξετάσουμε τόσο τις ε, τροπολογίες όσο και τις ε, συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.